Τώρα το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Ο κύριος Λόπες Γαρίγα, του Συμβουλίου, έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. πρόκειται για ένα θέμα ζωτική σημασία για το Συμβούλιο και για την Ισπανική Προεδρία. Είναι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 για την ανάπτυξη και την απασχόληση ποιότητας. Το είπαμε και νωρίτερα ότι βγαίνουμε από την χειρότερη οικονομική κρίση μετά τη δεκαετία του 30 και πρέπει να φροντίσουμε η ανάκαμψη αυτή που ξεκινάει που αρχίζει και εμφανίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τις προβλέψεις που παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να φροντίσουμε αυτή να συνεχιστεί και συγχρόνως να περιορίσουμε τις κοινωνικές συνέπειες της κρίσης. Επιπλέον όμως πρέπει πρόθεσμα... να δούμε τι κάνουν τα κράτη-μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά και να κοιτάξουμε και λίγο πιο μακριά στα τέλη της δεκαετίας της επόμενης και να φροντίσουμε για το σωστό κοινωνικό μοντέλο στην Ευρώπη. Αυτή είναι η δυτή πρόκληση που περιλαμβάνεται στην στρατηγική μας 2020. Θέλουμε δηλαδή να μην περάσουμε ξανά από μια τέτοια κρίση και θέλουμε να φροντίσουμε να γίνει αυτό με μια στρατηγική ανάπτυξης, με ένα αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο να είναι καλά προσαρμοσμένο στους καιρούς που ζούμε και επιπλέον έχουμε μια στρατηγική ανάπτυξης πραγματική και απαιτητική. Αυτή είναι η πρόκληση, πολιτική και οικονομική, που θα αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η στρατηγική 2020 ξεκίνησε να συζητιέται σε επίπεδο ηγετών κρατών και κυβερνήσεων στις 11 Φεβρουαρίου άτυπα. Μετά και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου συζήτησε για αυτήν και συζητιέται και σε πολλές ομάδες στο Συμβούλιο υπό Ισπανική Προεδρία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου ενέκρινε την στρατηγική 2020 που οριστικά θα εγκριθεί στο Συμβούλιο του Ιουνίου και εντόπισε τα στοιχεία, τη δομή, ακόμα και τον οδικό χάρτη για το μέλλον της στρατηγικής αυτής. Πρόκειται για την γνώση και την καινοτομία, την αηφόρα οικονομία, βιώσιμη οικονομία, αλλά μιλήσαμε και για το κοινωνικό μοντέλο και την απασχόληση. Πρόκειται για στόχους κλειδί που έχουν ήδη ποσοτική έκφραση όσον αφορά για την απασχόληση, την ανεργία, όταν πρόκειται για το ποσοστό του ΑΕΠ που θα πηγαίνει στην έρευνα και την καινοτομία, για το κλίμα με το 2020. αλλά μένει και το θέμα της κατάρτισης και εκπαίδευσης, πράγματα τα οποία ακόμα δεν έχουν εκφραστεί ποσοτικά, όπως και η κοινωνική ένταξη και η απάλληψη της ένδυας. Όλα αυτά βέβαια βάσει της ανακοίνωσης που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που ήταν αποφασιστική σημασίας για την ε, απόφαση, τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Μάρτιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η δομή τώρα της στρατηγικής 2020. Πρώτον, κατευθυντήριες γραμμές. Η πρόταση έγινε για κατευθυντήριες γραμμές, για προσανατολισμούς. Θελήσαμε να συζητήσουμε προκειμένου το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ και το Συμβούλιο τον Ιούνιο να αποφασίσει με τη σύμφωνη γνώμη βέβαια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία απαιτείται. Δεύτερον, έχουμε τους βασικούς στόχους, στους οποίους αναφέρθηκα πριν. Και τρίτον, υπάρχει και μια καινοτομία της νέας στρατηγικής, που είναι η εθνική στόχη. Κάθε κράτος πρέπει να θέσει τους εθνικούς του στόχους, που βέβαια να συμπεριλαμβάνονται και στους ευρωπαϊκούς στόχους και να στηρίζονται από την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Μιλήσαμε επίσης για τα μποτελιαρίσματα που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο η Ισπανική Προεδρία θα επικεντρωθεί στα προβλήματα εκείνα που έχουν κυρίως να κάνουν με την εσωτερική αγορά. Επιτέχουμε τις πρωτοβουλίες, τις ε, μεγάλες πρωτοβουλίες που έχουν ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρώτη και κύρια υπό Ισπανική Προεδρία ήδη έχουμε την ψηφιακή ατζέντα που τον Μάιο θα συζητηθεί στο Συμβούλιο μετά από μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την οποία μας υποσχέθηκε για τις 18 Μαΐου. Τέλος, κυρία Πρόεδρε, θα έχουμε και ειδικέ συζητήσεις για τη στρατηγική αυτή στο Συμβούλιο, σε διάφορες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου και θέλουμε οι συζητήσεις αυτές να γίνονται δημόσια, για παράδειγμα στο επόμενο Συμβούλιο Εκπαίδευσης, την επόμενη εβδομάδα. Θα είναι ανοιχτή η συζήτηση. Βέβαια, οι εργασίες δεν θα ολοκληρωθούν τον Ιούνιο. Θα συνεχιστεί η ανάπτυξη της στρατηγικής 2020 που στη συνέχεια θα πρέπει να εφαρμοστεί και μέσω και των εθνικών προγραμμάτων. Και τέλος, το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι για την διακυβέρνηση της στρατηγικής θα μας απασχολήσει πολύ. Τόσο η Ισπανική Προεδρία όσο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ο πρόεδρος Φανρομπάη θα ασχοληθούν πολύ με τον προσανατολισμό της στρατηγικής αυτής, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα αποτελέσουν και τα δύο θεσμικά όργανα κλειδί για την εφαρμογή της στρατηγικής αυτής. Έχουμε ήδη αρκετά μέσα και όλοι έχουμε την βούληση να πετύχει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λόπες Γαέρο. Τώρα ο κύριος Μπαρόζο. Εκ το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αξιότιμα μέλη, η Ευρώπη πρέπει να πάρει αποφάσεις. Ε, μια ε, στεναρή ε, στάση απέναντι στις αγορές ή ως όσον ναι αυτό σωθεί το. Μεγαλύτερη συνεργασία ή μια κατάσταση που θα ζούσαμε δεκαετίε ολόκληρε, ε, όπως το παρελθόν. Τους τελευταίους μήνες είδαμε εξελίξεις που ήταν η πτυτικότητα των αγορών που δεν υποχωρούσε, ανάγκη για χρηματοοικονομικές μεταρρυθμίσεις, για εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών. Όλα αυτά ε, μας έκαναν να καταλάβουμε ότι η επιλογή είναι μία και σαφής. Θα πρέπει να τονίσουμε τη σημασία της ευρωπαϊκής διάστασης περισσότερο από ποτέ. Και τώρα έχουμε την ευκαιρία να το πράξουμε ακριβώς γύρω από αυτούς τους στόχους της ε, Ευρώπης 2020. Μου ζητήσατε να μιλήσω για το πακέτο αυτό. Κοιτάζοντας τα μέτρα για μια ε, ανάπτυξη ε, έξυπνη, ευφυή, αηφόρο, βιώσιμη, αυτά δεν θα πρέπει να τα βλέπουμε ξεκομμένα από την γενικότερη κατάσταση. Σήμερα ζούμε μια κρίση. Θα πρέπει όλοι μαζί να συνεργαζόμαστε σε όλους τους τομείς για να καλύψουμε τα κενά στα πλαίσια του κανονισμού και της εποπτείας των χρηματαγορών για να επανέλθει η μακροοικονομική ε, σταθερότητα και η υγιή οικονομικά να αρχίσουν οι μεταρρυθμίσεις ε, που να οδηγήσουν την Ευρώπη στο δρόμο της αηφόρου ανάπτυξης και των ε, θέσεων απασχόλησης. Και αυτές οι πτυχές όλες εξίσου ισχύουν και είναι σημαντικές αν θέλουμε να φτάσουμε στους στόχους μας. Χρειάζεται λοιπόν μια συνολική, μια καθολική προσέγγιση, μεταρρύθμιση των χρηματαγορών, ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης, μια Ευρώπη βιώσιμη, με αηφορία, με συμπερίληψη, με ε, το G20 επίσης, γιατί πολλά θέματα έχουν και εξωτερική διάσταση. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ό,τι έχουμε στη διάθεσή μας ως μέσο και ως μέτρο και ως επίπεδο για να επηρεάσουμε ε, ε, όλα τα άλλα σύντομα να αναφερθώ, δεν θα επανέλθω στα χρηματοοικονομικά που ανέφερα στην προηγούμενη μου δήλωση. Επιτρέψτε μου να σας αναφέρω την ομάδα των 20, το G20. Χρειάστηκε να βελτιώσει την οικονομική διακυβέρνηση ε, παγκοσμίω. Ε, θα πρέπει ε, τώρα να δοθεί μια νέα όθηση με νέες ιδέες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συνεισφέρει στην κατάσταση αυτή έτσι ώστε ε, και τα συμφέροντα και τα ενδιαφέροντα και των 27 κρατών μελών να αντανακλώνται στην εργασία μας. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει τον Ιούνιο στο Τορόντο και στη Σεούλ την ηγετική της ε, θέση και να στείλουμε ένα σαφέ μήνυμα από του G20 για τη στρατηγική εξόδου και υποστήριξη τη ανάκαμψη της οικονομίας. Όλες οι μεγάλες οικονομίες θα πρέπει να παίξουν το ρόλο τους και παγκόσμια να αντιμετωπίσουμε κάποιες από τις ανισορροπίες που πραγματικά είναι ε, στην πηγή της κρίσης. Θα πρέπει επίσης να βεβαιωθούμε ότι θα μοιραστούν όλα τα μέλη του G20 το βάρος, το ε, άχθος της ανάκαμψης της οικονομίας θα πρέπει να ενισχυθεί γενικότερα η οικονομική συνεργασία στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό εδώ. Έχει σημασία η Ευρώπη να έχει συντονισμένη προσέγγιση στη G20. Άλλος στόχο είναι η μεταρρύθμιση των χρηματαγορών, να διατηρήσουμε την πίεση στους ε, διεθνεί εταίρου μα να ε, μας δίνουν εγκαίρως ε, στοιχεία και να εφαρμόζουν τους κανόνες που ήδη υπάρχουν για ίσους κανόνες παιχνιδιού. Σχηρό μήνυμα πρέπει να σταλεί για το πώς μπορεί ο χρηματοοικονομικός τομέα να συνεισφέρει στη ε, χρηματοδότηση της ανάκαμψης. Μια συντονισμένη προσπάθεια χρειάζεται, μια παγκόσμια συμφωνία για ε, τις τράπεζες, για τη σταθερότητά τους αυτό θα μπορούσε να συμπληρωθεί και από ένα τέλος χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων ή κερδών. Αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολη συζήτηση, το ομολογώ. Ήδη προκατακτικά το συζητούμε στο G20, αλλά πολύ είναι αντίθετη με την ιδέα αυτή. Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να τη συνεχίσουμε. Το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πιο ισχυρό σίγουρα αν μιλήσουμε με μία φωνή και μπορούμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει τη δική της δουλειά. Γι' αυτό θα πρέπει να στοχεύουμε να έχουμε συμφωνία για τον κανονισμό για τις βασικές χρηματοοικονομικές ε, υπηρεσίες που σας ανέφερα προηγουμένως. Χρειάζεται ευελιξία και ρεαλισμός από το Κοινοβούλιο αλλά και από το Συμβούλιο. Και έρχομαι τώρα στη Συμφωνία του 2020 στη μερίσια διάταξη ε, ως τμήμα αυτής της καθολικής προσπάθειας που σας είπα. Όπως γνωρίζετε, πολλά στοιχεία από τη στρατηγική του 2020 εγκρίθηκαν το Μάρτιο από αρχηγούς ε, κρατών και κυβερνήσεων. Είχαμε επανειλημμένα την ευκαιρία στο Κοινοβούλιο σας να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, ακόμα και πριν κάνουμε την πρόταση, ε, σας συμβουλευτήκαμε. Και τώρα θα πρέπει να καθορίσουμε τη στρατηγική μας, ε, έτσι να δώσουμε σάρκα και οσά στις λεπτομέρειες. Είναι κατεπίγουσα η ανάγκη για δράση. Αυτό το έχουμε καταλάβει όλοι περισσότερο από ποτέ. Δεν θέλω να επαναλάβω την προηγούμενη συζήτηση, αλλά ε, αυτή η χρηματοοικονομική κρίση και τα προβλήματα της Ευρωζώνης κατέδειξε ότι θα πρέπει να κάνουμε βαθύτερες μεταρρυθμίσεις με τρόπο συντονισμένο και αποφασιστικό. Καλύτερος λοιπόν συντονισμός των οικονομικών μας πολιτικών είναι η καρδιά ίδια της Ευρώπης για το 2020 και πριν την ελληνική κρίση. Κάναμε προτάσεις, ε, δίναμε ιδέες για περισσότερο συντονισμό της οικονομικής πολιτικής. Αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε, είναι απαραίτητο για να αποφευθεί μελλοντική κρίση να ε, επανακάμψει η οικονομία και η ανάπτυξη με καλύτερες και περισσότερες θέσεις απασχόλησης και τελικά ε, ένα βιώσιμο αηφόρο ε, μέλλον για την Ευρώπη. Πέντε είναι οι στόχοι που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μεγάλη η συνένεση. Έχουν δοθεί και αριθμητικά στοιχεία για την απασχόληση, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την έρευνα και την ανάπτυξη. Για την εκπαίδευση τώρα Θέλουμε να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών που εγκαταλείπουν νωρί το σχολείο, να αυξηθεί ο αριθμό των πτυχιούχων τριτοβάθμια εκπαίδευση ή αντιστοίχων. Ε, αυτό θα το εγκρίνει το Συμβούλιο τον Ιούνιο με βάσει την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση, θέλω αριθμητικό στόχο για την καταπολέμηση τη φτώχεια και του κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε ε, το σκάνδαλο αυτό το συνεχέ με κίνδυνο 80 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτε να πέσουν στη φτώχεια. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να πείσω τα κράτη-μέλη για τη σημασία του στόχου αυτού. Γνωρίζω ότι το Κοινοβούλιο συμμερίζεται την αποφασιστικότητά μα. Ευρώπη 20 2020 θα πρέπει να είναι ισορροπημένη και βεβαίω δεν μπορεί να νοείται κοινωνική ισότητα χωρί ανταγωνιστική αγορά. Μια Ευρώπη οικονομικά ανταγωνιστική όμω θα πρέπει να συνοδεύεται και από κοινωνική δικαιοσύνη. Οι εθνικοί στόχοι θα επιτρέψουν καλύτερη και αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και έλεγχο των κρατών μελών για να φτάσουμε στου στόχου μα. Τα κράτη-μέλη είναι στη διαδικασία τώρα ε, ε, θέσης αυτών των στόχων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω να ε, αρχίζουν αυτά να εφαρμόζονται το σύντομότερο. Την περασμένη εβδομάδα κάναμε μία πρόταση για τις κατευθυντήριες γραμμές και για τη στρατηγική για το 2020. Είναι πιο περιορισμένος ο αριθμός των ε, κατευθυντήριων γραμμών, 10 πλέον ε, σε αντίθεση με 24 που είχαμε, για να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει περί τίνος πρόκειται να το εστερνιστεί. Είναι πρόοδος. Τον Ιούνιο το Συμβούλιο θα πρέπει να δώσει την έγκρισή του ε, βεβαίως για τις κατευθυντήριες γραμμές, αλλά βεβαίως θα εγκριθεί μόνο εφόσον το έχουμε συζητήσει μαζί σας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζω αυτό να γίνει το συντομότερο. Κυρίες και κύριοι, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Η στρατηγική 2020 για την Ευρώπη δεν είναι απλώς μια έμπνευση, ένα ευχολόγιο, ε, μια απαρίθμηση στόχων, ένα όραμα. Είναι ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων θα αναλυφθεί η δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να γίνουν σε κάθε μία από τις 27 χώρες. Σε κάθε μία χώρα. Ε, σε πλήρη σεβασμό του, ε, της επικουρικότητας. Να ξέρουμε τι πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τι σε εθνικό. Και κλειδί εδώ είναι η εφαρμογή. Όπως είπε ο αξιότιμος εκπρόσωπος του Συμβουλίου κύριος Λόπες Γκαρίντο, Σήμερα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επίγνωση στα κράτη-μέλη της ανάγκης ε, της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Ελπίζω τα κράτη-μέλη να έχουν διδαχθεί ε, από τις ε, ελλείψεις και αδυναμίες της ε, στρατηγικής της Λισαβόνας. Πολλοί από τους στόχους ήταν καλοί, όχι όλοι, αλλά δεν υπήρξε αρκετή υιοθέτηση των στόχων και αρκετό σθένος στην εφαρμογή των προγραμμάτων. Δεν τα εστερνίστηκαν. Γι' αυτό θα πρέπει να κλείσει αυτό το έλλειμμα, αυτό το χάσμα στη στρατιστική της Λισαβόνας. Εκεί έχετε εσείς να διαδραματίσετε ένα κρίσιμο ρόλο για την επιτυχία της στρατηγικής 2020. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτός από συνομοθέτης μπορεί να κινητοποιεί και τους πολίτες με τρόπο πολύ αποτελεσματικό. Και γιατί όχι, επίσης και τα εθνικά κοινοβούλια, επίσης είναι πολύ κρίσιμο, πολύ σημαντικό. Αν μου επιτρέπετε να σας αναφέρω, να έχετε καλές σχέσεις, δεσμούς με τα εθνικά κοινοβούλια, έτσι ώστε να βεβαιωθείτε ότι ε, δεν θεωρούνται οι μεταρρυθμίσεις αυτές ως μεταρρυθμίσεις που κάνουν οι Βρυξέλλες ή επιβάλλουν κάποιοι από τις Βρυξέλλες ή από το Στρασβούργο, αλλά παντού σε όλα τα επίπεδα των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Είναι επίγουσα ανάγκη για μεταρρυθμίσεις και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι φορείς, κοινωνική, οικονομική και πολιτική, σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης, αλλά και οι κοινωνικοί εταίροι. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Καλωσορίζω όλες τις ανακοινώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργό κ. Σαπατέρο για τη συμπερίληψη και των κοινωνικών εταίρων. Και θα πρέπει να υπάρξει κοινή διακυβέρνηση με κοινό συντονισμό. Όλα τα εργαλεία που έχουμε και ε, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και η Στρατηγική 2020, όλα αυτά ταυτόχρονα να υλοποιούνται για να φτάσουμε στους στόχους μας. Για ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Μελέτης του Συστημικού Κινδύνου για μεταρρυθμίσεις, για ανταγωνιστικότητα, ε, μακροοικονομικές εξελίξεις. Όλα αυτά θα μας φέρουν ε, έξω από την κρίση σε μια ευφυή, βιώσιμη και φόρο ανάπτυξη. Αυτός είναι ο δρόμος. Ο μόνος δρόμος δεν μπορούμε σοβαρά να μιλάμε για οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διαχωρίσουμε τη μακροοικονομία από τη μικροοικονομία, τα εσωτερικά μας από τα εξωτερικά. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, όλη την ενέργειά μας ε, μια καθολική συνολική προσέγγιση, μόνο έτσι θα ε, προχωρήσουμε και θα δώσουμε και κάποια αξιοπιστία και εμπιστοσύνη στη στρατηγική μας. Μίλησα για μια δύσκολη επιλογή ε, και γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τι θα διαλέξει. Είμαι πεπισμένος ότι και εσείς είστε στο πλευρό μας υπέρ της Ευρώπης αποφασιστικά και υπολογίζω στην υποστήριξή σας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρους των πολιτικών ομάδων τώρα το λόγο έχει η κυρία Βόρτμαν Κόλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Πρόεδρε Μπαρόσο, αγαπητέ Υπουργέ, η συζήτηση αυτή για τη στρατηγική 2020, σωστά, πρέπει να προχωρήσει και έχει άμεση σχέση και γι' αυτό και ακολούθησε τη συζήτηση που κάναμε για την οικονομική κρίση. Γιατί πραγματικά πρόκειται για το θέμα η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση μπορεί να ενισχύσει και την οικονομική διακυβέρνηση. Μιλάμε και για την οικονομική πολιτική, όμως το κύριο πρόβλημα είναι ότι ένα κράτος μέλος ακύρωσε τελικά τις δεσμεύσεις του. Δεν γίνεται όμως, γιατί τα χρήματα για τη σταθερότητα και για την ανάπτυξη πρέπει εκεί να πηγαίνουν. Αυτό είναι το μάθημα που πρέπει να πάρουμε. Και αυτό είναι που πρέπει να μας βοηθήσει να χαράξουμε τη στρατηγική μας για το 2020. Η ομάδα μας θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι φιλόδοξη όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση και να αποτελεί σε αυτή μέρος της στρατηγικής 2020. Και από το Συμβούλιο περιμένουμε να πάρει φιλόδοξες αποφάσεις, να βάλει φιλόδοξους στόχους για τα κράτη-μέλη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν χρειαστεί, θα το απαιτήσει αυτό. Τα επόμενα χρόνια λοιπόν πρέπει να φροντίσετε αυτά τα θέματα να συμπεριληφθούν στη στρατηγική 2020. Και αυτό προς το συμφέρον της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, υπέρ της απασχόλησης και των πολιτών μας. Οι αναταραχές στην Ευρωζώνη, Πρόεδρε, έδειξαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε υγιή δημοσιονομικά, για τη σταθερότητα του ευρώ, για την οικονομική σταθερότητα, αλλά και για να προλάβουμε να πληρώσουν την ύφη επόμενε γενιές, τα παιδιά μας. Η μεταρρύθμιση, η μεταρρύθμιση των δημοσιονομικών λοιπόν αποτελεί προϋπόθεση για να πετύχει η στρατηγική μας για το 2020 και για να έχουμε ανάκαμψη στην οικονομία. Και γι' αυτό και είναι τόσο σημαντικό, Επίτροπε Ρεν, να έρθετε με προτάσεις ώστε να ενισχυθεί το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Να υπάρχουν οι προληπτικοί μηχανισμοί και να ελέγχονται καλύτερα τα δημοσιονομικά στις χώρες μέλη. Θέλω να σας ενθαρρύνω λοιπόν, η ομάδα μας ολόκληρη, ώστε να αναλάβετε ως Επιτροπή την ευθύνη και να έρθετε με ένα φιλόδοξο σχέδιο. Να μας στηρίξετε και εμείς θα στηρίξουμε ένα τέτοιο φιλόδοξο σχέδιο. Το Συμβούλιο με την Επιτροπή επίσης πρέπει να φροντίσει να γίνει αυτή η δουλειά να στηριχθεί και να ενισχυθεί το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξη Το Συμβούλιο είναι καλό που έφτιαξε μια task force Ελπίζω όμως ότι το Συμβούλιο μέχρι τα τέλη της χρονιάς θα μπορέσει να στηρίξει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόεδρε, οι δυνατότητε που δίνει η συνθήκη τη Λισαβόνα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πλήρω υπέρ τη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, να ενισχυθεί αυτή. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η ε, κυρία Μπερέ για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε της ε, Κομισιόν, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Η σύνδεση ανάμεσα στις δύο συζητήσεις που είχαμε είναι πνευματικός ε, συνεπής. Τώρα αν μεταφράζεται στην πράξη έχουμε αμφιβολίες στο πλαίσιο της Σοσιαλιστικής και Δημοκρατικής Ομάδας γιατί όταν βλέπει κανείς το κείμενο όπως μας προτάθηκε από την Κομισιόν και μέσα στο πλαίσιο μια στρατηγική εταιρική σχέση θέλετε να υιοθετήσετε τον Ιούλιο χωρί το Κοινοβούλιο να μπορεί να εκφραστεί για τι κατευθυντήριε γραμμέ για την απασχόληση με ρητό τρόπο, ε, δεν βλέπουμε πού βρίσκεται η συνοχή. Πώ ε, μπορείτε να φανταστείτε ότι θα δεσμευτούμε για τα επόμενα 10 χρόνια χωρίς να κάνουμε έναν απολογισμό του τι ήταν και τι έκανε η στρατηγική της Λισαβόνας. Μας λέτε ότι όλα άλλαξαν και ότι δεν έχουμε πια 27 κατευθύνες γραμμές, έχουμε 10. Μα αυτή είναι η αλλαγή μόνο, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής. Η συνοχή είναι ότι αν θέλουμε να επιτύχουμε τη στρατηγική του 2020 πρέπει να ξεκινήσουμε από το σημείο που βρισκόμαστε πριν να δούμε πού κατευθυνόμαστε. Πρέπει να δούμε δηλαδή να βάλουμε στόχους, να δούμε πού θέλουμε να πάμε, να φτάσουμε. Εδώ που βρισκόμαστε σήμερα είμαστε στην πιο σημαντική κρίση που έχει ποτέ γνωρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη από τη δημιουργία της. Σοβαρότερη κρίση δεν έχει υπάρξει. Αυτό δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα σε μια στρατηγική εξόδου από την κρίση ε, που θα ήταν ε, το αίτημα της ε, διαφυγής το δημόσιο τομέα για να φύ, από τις ευθύνες του ώστε να αφήσουμε ελεύθερο το πεδίο για τις ε, δυνάμεις της αγοράς. Ξέρετε πολύ καλά κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής ότι δεν είμαστε και τόσο πλούσιοι. Έχουμε ένα εργαλείο που λέγεται Σύμφωνο Σταθερότητας. Έχουμε και άλλα που ονομάζονται δημοσιονομικές προπτικές. Αν δεν συνδεθούν μεταξύ τους όλα αυτά ξεκάθαρα δεν θα φτάσουμε πουθενά. Και επιτά, όταν βλέπουμε από πού ξεκινάμε Έχουμε λόγους για ανησυχία. Καταρχήν εμείς οι σοσιαλιστές δημοκράτες ζητάμε κατεπηγόντως τα κράτη να μην υπόκειται πλέον στην κερδοσκοπία των αγορών. Και δεν είναι θέμα της Ελλάδας ή του ενός ή του τάδε ή κράτους μέλου. Είναι θέμα του παιχνιδιού του ντόμινου και του ελεύθερου πεδίου στην κερδοσκοπία. Και γι' αυτό και προτείνουμε τη δημιουργία ενός μηχανισμού οικονομικής σταθερότητας που θα επιτρέψει να προστατευτούν τα κράτη-μέλη από αυτή την κερδοσκοπία, ώστε να κάνουν αυτό που οφείλουν να κάνουν. Δηλαδή να ξαναβρούν το δρόμο της ανάκαμψης που θα επιτρέψει να διασφαλιστεί και το κοινωνικό μοντέλο. Γιατί όλοι το γνωρίζουν και όλοι το έπανε στη διάρκεια αυτή της κρίσης ότι το κοινωνικό μας μοντέλο είναι το καλύτερό μας εργαλείο, η δύναμή μας για την παγκοσμιοποίηση. Και αν η στατικική σημαίνει περικοπές δημοσιονομικές που σκοτώνουν αυτό το κοινωνικό μοντέλο, η Ευρώπη αύριο θα ιτηθεί στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού και οι ικανότητέ τη να υποστηρίξει αυτό το μοντέλο το οποίο εμεί αντιπροσωπεύουμε, το, θα χαθεί ο αγώνα και θα αφήσουμε τον χώρο για τι άλλε υπήρου, εκτό και αν βέβαια θα αφήσουμε το θέμα μόνο στο παιχνίδι των αγορών. δεν είναι αυτό να μας για το μέλλον. Η κυρία Εκ τώρα για τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ. Γνωρίζουμε εδώ και πολλού μήνε πω η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. ξέρουμε πω το ευρώ. Ε, ε, ε, χάνει την αξία του και κανένας δεν αφισβητεί πως η Ευρώπη διανύει μια πολύ σοβαρή κρίση και μόλις ε, νομίζαμε ότι θα είχαμε πάλι ορθοποδήσει βλέπουμε ότι έχουμε πρόβλημα ανταγωνιστικότητας, παραγωγικότητας και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ωστόσο εξακολουθούν να τσακώνονται ε, να λογομαθούν για το τι χρειάζεται να κάνουν. Ε, τέρμα τα λόγια, χρειάζεται δράση τώρα. Χρειαζόμαστε δεσμευτικούς στόχους, νέα διαφανή μέτρα για τον έλεγχο των εκθέσεων για κάθε κράτος μέλος. Χρειάζεται θεμελιώδη σεβασμό στους συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης και χρειάζεται Χρειάζονται αξιόπιστα και αληθινά στοιχεία επί των οποίων να βασίσουμε τι αποφάσει μα. Πρέπει επιπλέον να πιέσουμε τι κυβερνήσει. Τα διευθυντικά ταμεία και άλλη ευρωπαϊκή στήριξη θα πρέπει να, να συνδέεται με την δυνατότητα τη κυβέρνηση κάθε φορά να μα δώσει σωστά στοιχεία. Και να κάνω μια σύγκριση. Όταν ένα μικρό ε, αγρότη κάνει λάθο μισό εκτάριο, χάνει την στήριξή του. Για όλα όσα κάνει για πολλά χρόνια. Αυτό το είδος την πρόταση πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό είμαστε και τόσο αυστηροί όσον αφορά τη διακυβέρνηση στο ψήφισμά μας το κοινο, το βουλε, το, του Κοινοβουλίου. Επίσης είναι πολύ απογοητευτικό που η Κομισιόν δεν κάνει προτάσεις που τις συζητάμε εδώ και χρόνια να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα για τη μελλοντική ανάπτυξη και μια στρατηγική ατζέντα θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη στρατηγική για το 2020. Να δώσω κάποια παραδείγματα. Διαπραγματευτήκαμε ένα σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης, ανάκαμψης. Το μεγαλύτερο τμήμα του δεν έχει επιβληθεί. Το Κοινοβούλιο ζήτησε να υπάρχει ένα δεύτερο πλάνο υπαναχώρησης που να συμπεριλαμβάνεται στα αποτελέσματα και δεν έχει ακόμα αυτό τεθεί σε εφαρμογή αποφασίσαμε σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο για νέα ενέργεια και τεχνολογία. Ακόμα είμαστε 50% πίσω στη χρηματοδότηση αυτού του στρατηγικού εργαλείου και το πιο αποτελεσματικό μέσο για να περιοριστούν οι εκπομπές των ε, αερίων του θερμοκηπίου είναι να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα στην ενέργεια, ε, την ενεργειακή αποδοτικότητα και αυτό θα πρέπει να μπει πάνω πάνω στην ημερήσια διάταξη για δράση. Αποτελεσματική νομοθεσία θα πρέπει πρέπει να αναβαθμιστεί γιατί δεν αποδίδει και χρειάζεται και το πρόγραμμα δράσης για την, αποδοτικό, την ενεργειακή αποδοτικότητα. Χρειάζονται ε, υποδομές για την ενέργεια χρειάζονται οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι της ενέργειας για να τους πούμε έτσι. Πρέπει να διασφαλίσουμε την τεχνική καινοτομία και επίσης χρειάζεται να ενθαρρύνουμε και να προωθήσουμε τη στρατηγική για τον αποκλεισμό της κοινωνικής, του κοινωνικού αποκλεισμού και την ένταξη των δύο φύλων. Υπό το φως αυτής της κρίσης θα πρέπει η ευθύνη, η Κομισιόν συγγνώμη, να σταθεί ε, στο ύψος ε, των περιστάσεων και να αναλάβει τις ευθύνες της και το, και το Συμβούλιο να γίνει πιο στεναρό, πιο δυνατό και να σταματήσει τις κοκορομαχίες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χάρμς για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι συνάδελφοι. Νομίζω φτάνουμε λίγο στην πολιτική πρόκληση, στην πολιτική προβοκάτσια το πρόγραμμα 2020 να θεωρείται ως η μεγάλη πρόκληση για την έξοδο από την κρίση. Αρκεί κανείς να δει την πολιτική μέχρι τώρα για τη ρύθμιση των χρηματαγορών. Και αν είμαστε και στοιχειοδός ειλικρινείς, θα πρέπει να πούμε ότι εδώ και μήνες, για να μην πω χρόνια, τάζουμε ε, ότι αυτές οι αγορές που είναι ασίδωτες θα ρυθμιστούν. Αλλά μέχρι τώρα έχουμε κάνει βηματάκια, νάνου, για να προχωρήσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Και ορίστε, η Ελλάδα μας δείχνει τι κάναμε. Σε αυτή την κρίση αποδεικνύεται ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα αρκετό. Οι πολίτες ε, ζήσανε αυτό που είπαμε εμείς ότι θα σώσουμε τις τράπεζες, δεν πειράζει, σφίξαν τα δόντια και το δεχτήκανε. Αλλά τώρα έρχονται να πληρώσουν τα σπασμένα. Και οι κρατικοί προπολογισμοί έχουν ήδη υπερφορτωθεί ε, για τις τράπεζες. Τώρα σώζουμε την Ελλάδα, είμαστε υποχρεωμένοι, δεν χωράει καμία αμφιβολία, πρέπει να το κάνουμε. Αλλά αυτό είναι και επιπλέον επιβάρηση των κρατικών προϋπολογισμών σε πολλά κράτη της Ένωσης. Οι τράπεζες είναι κερδοφόρες και χειροκροτούμε όταν λέμε ότι συμμετέχουμε Λένε αυτέ, ε, θα μπούμε λίγο εθελοντικά να βοηθήσουμε την Ελλάδα κι εμεί. Ποιο οι κερδοφόρε τράπεζε και εμεί χειροκροτούμε. Κύριε Μπαρόζο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια αγορά που συμμετέχουν 27 χώρες. Θα πρέπει να βάλετε ένα φόρο, ένα τέλος χρηματικών συναλλαγών, δεν ξέρω τι θα βρείτε, ε, έτσι ώστε να μετριαστεί η πείνα των κερδοσκόπων. Χρειαζόμαστε ένα εργαλείο πραγματικά για να μπορούμε να είμαστε και δίκαιοι και αυτοί που κερδοσκοπούν και κερδίζουν από τις επιθέσεις στο ευρώ θα πρέπει να πληρώνουν. Γιατί από τους κρατικούς προϋπολογισμούς δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο που ξεκινήσαμε να συνεχίσουμε. Και σε αυτό το έγγραφο που μας δώσατε μου λείπει ακόμα αυτό το όραμα της μελλοντική πορείας. Και γνωρίζω ότι ε, χρειάζεται λέτε αυτό να γίνει παγκοσμίω από το κλίμα μας λέτε ότι είναι παγκόσμια η πρόκληση και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Κλιματική αλλαγή λοιπόν και άλλη κρίση που δεν βγαίνουμε καθόλου παρά μόνο βυθιζόμαστε όλο και πιο βαθιά γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε τα σωστά βήματα. Είναι πραγματικά αξιοθρύνητο το γεγονός ότι ε, σήμερα λίγο πριν τη συζήτηση αυτή είδαμε ότι η Κόνη Χέντεγκαρτ δουλεύει σαν τυφλοπόντικας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσπαθεί τον ελάχιστο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τον περάσει. Και αν δούμε την ε, σημερινή κατάσταση, νομίζω θα πρέπει οπωσδήποτε να αυξήσουμε τους στόχους στο 30%. Είναι απαραίτητο. Το περίφημο εμπόριο εκπομπών ρήπων στην Ένωση, αν δεν αυξηθεί ο στόχος δεν μπορούμε ε, ούτε τέτοιο να έχουμε. Ε, εμπόριο. Γιατί αν το διοξίδιο του άνθρακα δεν ε, έχει την τιμή που πρέπει, αν οι στόχοι μας δεν είναι αρκετά φιλόδοξοι, τότε συζητάμε χρόνια ολόκληρα, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας και ε, απεμπολούμε και τον ίδιο μας το στόχο. θα πρέπει να μετασχηματιστεί η ευρωπαϊκή ε, οικονομία προς μια βιωσιμότητα, προς μια εφορία. Τα βάζετε και στις επικεφαλίδες των προγραμμάτων σας. Όλοι συμφωνούν και χαροπά συνεργάζονται. Αλλά η δική σας Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Μπαρόσο, δεν μας είπε τι θα το κάνει αυτό το πρόγραμμα και πώς θα εφαρμοστούν οι στόχοι στην ευρωπαϊκή οικονομία. Με ποια μέσα, με ποια εργαλεία, με ποια κίνητρα θα γίνουν όλα αυτά. Η κυρία Εκ έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα σε επιμέρους τομείς. Νομίζω ότι χρειάζεται πολλή δουλειά το πρόγραμμά σας αυτό και μέχρι τώρα αυτά που έχουμε στα χέρια μας δεν νομίζω ε, ότι μπορεί να κάνει το κοινοβούλιο να πει ότι μετά τη Λισαβόνα είναι αυτή η νέα σπουδαία πορεία, η νέα σπουδαία κίνηση. Από την αποτυχία της ε, στρατηγικής Λισαβόνας έχουμε τώρα την επόμενη αποτυχία του 2020. Ευχαριστώ κύριο Καμίνσκι για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, Νομίζω πως ε, σήμερα έχω ένα από τα πιο δύσκολα έργα. Ε, ο κύριος Μπαρόζο επίσης έχει πολύ δύσκολο έργο. Ε, πρέπει να πείσει την αριστερά και τη δεξιά για το βάσιμο των προτάσεών του και να μπορέσει να πλεύσει ανάμεσα από όλες αυτές τις προτάσεις. Η πρόταση για το 2020 ε, ε, είναι εξαιρετική. Πραγματικά εγώ εντυπωσιάζομαι όταν ακούμε εδώ ε, μέσα στην αίθουσα διάφορα που, που διάφορους που λένε ότι για να βελτιωθεί η κατάσταση που είναι πολύ δύσκολη σήμερα θα χρειαστούν πολύ, πολλές προσπάθειες. Εγώ 18 χρόνια της ζωής μου τα πέρασα στην ε, λαϊκή δημοκρατία της Πολωνίας. Εσωτερικό εμπόριο μόνο υπήρχε ε, και υπήρχε ένας υπουργός αλλά δεν υπήρχε εσωτερικό εμπόριο καν. Ε, σήμερα εδώ και 20 χρόνια ευτυχώς δόξα σε Θεός δεν έχουμε πλέον υπουργό εσωτερικού εμπορίου αλλά έχουμε εσωτερικό εμπόριο Πραγματικά η λύση δεν είναι περισσότερε ρυθμίσει, δεν είναι περισσότερε φόροι, δεν είναι περισσότερη παρέμβαση. Είναι σαφέ ότι είμαι από αυτού που είναι υπέρ του ελεύθερου εμπορίου. Πιστεύω πω ο ρόλο του κράτου είναι σημαντικό για να ρυθμιστεί η αγορά, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην χρήση τέτοιων ε, μέσων. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι αν θέλουμε να είμαστε έντιμοι και να μιλήσουμε για την ανάπτυξη στην Ευρώπη, να θυμηθούμε κάποια στιγμή την νομοθεσία, α πούμε, την οδηγία για τις υπηρεσίες. Σκεφτείτε τι συνέβη με εκείνη την οδηγία, εδώ σε αυτό το σώμα. οι τρεις χωρίς τις τρεις ελευθερίες των υπηρεσιών, των κεφαλαίων και των ανθρώπων η Ευρώπη δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Και εδώ ακούμε σήμερα πως δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε με άλλους πολιτικούς, οικονομικούς χώρους όσον αφορά την ολοκλήρωση. Μα εμείς έχουμε υπερβολικά πολλούς κανόνες, υπερβολικά με πολλή νομοθεσία και τελικά καταλήγουμε στο να σπρώχνουμε την ανταγωνιστικότητα της υπήρου μας προς άλλες υπήρους θα πρέπει αυτό να το ελέγξουμε και πρέπει να βρούμε από την κρίση. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως πρέπει να βοηθήσουμε την Ελλάδα γιατί για μας, τους Πολωνούς, η λέξη αλληλεγγύη έχει τεράστια σημασία. Πρέπει να δείξουμε σήμερα πως έχουμε αλληλεγγύη με την Ελλάδα και δεν έχω αμφιβολία καμία από αυτό. Θέλω να επαναλάβω πως πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε η Ευρώπη να βγει από την οικονομική κρίση. Γιατί δεν είναι μόνο το πρόβλημα εκατομμυρίων οικογενειών, αλλά είναι και το πρόβλημα της πίστης στο μέλλον μας. Πρέπει να πιστεύουμε στην επιτυχία μας και εγώ το πιστεύω αυτό. Ευχαριστώ. Ε, το λόγο έχει τώρα η κυρία Ζήμερ για 1,5 λεπτό. Ακούω τη συζήτηση για το τελευταίο θέμα και τη σκέφτομαι και τη συζήτηση που κάνουμε τώρα και τη συγκρίνω. Από ό,τι φαίνεται ε, ε, μιλάμε για δύο παράλληλους κόσμους. Από τη μια έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με χώρες όπως Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία σε απόλυτη κρίση και άλλες χώρες όπως η Γερμανία ή η Γαλλία να μπλοκάρουν και η άλλη συζήτηση μας δείχνει μια Ευρωπαϊκή Ένωση για την οποία αναπτύσσουμε μια στρατηγική που σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και στις προκλήσεις της. Ούτε με τη στρατηγική αυτή έχουμε ε, χαράξει νέο δρόμο για τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε απαντήσεις δίνουμε που να αντιμετωπίζουν τα μέσα και τα εργαλεία που δεν ε, λειτουργούν Πού είναι οι αρμοδιότητες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρατών μελών, ποια είναι η σχέση της Ευρωζώνης και των χωρών που δεν συμμετέχουν στην Ευρωζώνη αλλά είναι μέλη της Ένωσης. Όλα αυτά τα θέματα των τελευταίων ετών και της διαδικασίας της Λισαβόνας δεν τα έχουμε υιοθετήσει, δεν έχουμε δώσει απαντήσεις στραμμένες προς το μέλλον. Δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ε, τι πρέπει να γίνει, τι θέλουμε να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε τι να εξελιχθεί εν πάση περιπτώσει για να ξέρουμε πού το πάμε. Πού είναι η Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση Οικονομική, το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Δεν μπορούμε να υποκρινόμαστε ότι θα συνεχίσουμε τη στρατηγική μα όπω και στο παρελθόν. Είναι επίγον πριν συζητήσουμε για την υλοποίηση του 2020 να αφήσουμε τη στρατηγική, να πάρουμε περισσότερο χρόνο να, να αναβάλουμε τι αποφάσει, να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε, τι θα πρέπει να κάνουμε και η κοινωνία των πολιτών και τα εθνικά κοινοβούλια να συμμετέχουν πολύ πιο ενεργά από ό,τι μέχρι τώρα. Αλλιώς ε, ε, θα πάμε όπως είμαστε σούμπιτοι στην καταστροφή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπλουμ. you call me? Yes. Sorry, I didn't hear you. Uh, Μου δώσατε το λόγο. Συγγνώμη, δεν άκουσα. Δεν σας άκουσα. Ζητώ συγγνώμη που δεν σας άκουσα. Και είναι κρίμα που Έφυγε ο κύριο Κόνμπεντιτ από την αίθουσα γιατί θα είχε μάθει πολλά. Εγώ είμαι πεπισμένο ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε ε, και πολλά για το 2020 γιατί ελπίζω πω δεν θα είμαστε πια εδώ. Και η Σοβιετική Ένωση φαίνεται πολύ παρόμοια. Είναι κεντροποιημένη, διεφθαρμένη, αντιδημοκρατική και ανίκανη. Ε, καθοδηγείται από τις μεγάλες business και από τους ε, ε, χοντρουλούς γραφειοκράτες. Δηλα... Αναφερόμαστε στην υποτιθέμενη κλιματική αλλαγή. Οποτεδήποτε οι λαοί τη Ευρώπη έχουν την ευκαιρία ενό δημοψηφίσματο, το απορρίπτουν. Οι Βρετανοί φυσικά δεν είχαν καν την ευκαιρία να πούν τη γνώμη του χάρη στην εξαπάτηση των τριών κομμάτων που είχαν πρόσβαση στην τηλεοπτική συζήτηση στη χώρα μου που ε, προωθήθηκε από το πλήρως διεφθαρμένο τηλεοπτικό σύστημα που αποκαλείται BBC. Σύντομα οι υπόλοιπε μεσογειακές χώρες θα καταρρεύσουν όπως και η Ελλάδα και ε, το κύμα θα φτάσει και στις βόρειες ε, ευρωπαϊκές χώρες που θα πρέπει να σπηλυρώσουν την ύφη τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας θα μας καταβρίσουν αφού θα τους αφήσουμε να βγάλουν τη οφίδια από την τρύπα σε αυτή την ε, ε, κατάσταση στην οποία θα μπορούσαμε κάλλιστα να είχαμε αποφύγει. Ευχαριστούμε. Ο κ. Ομπερμάγερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε η ανάπτυξη η βιώσιμη και η μόνιμη, ναι, αυτά είναι μεγάλα λόγια. Αλλά εμένα με ανησυχεί το εξή. Οι νέε στρατηγικέ, η νέα στρατηγική δεν θα έχει την ίδια τύχη όπω και η προηγούμενη. Πώ οι περιφέρειε και οι Δήμοι θα εμπλακούν, ούτω ώστε αυτή η στρατηγική να είναι αποτελεσματική, πώ θα εξηγιανθούν οι εθνικοί προπολογισμοί. Και μέσα σε όλα αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να μην εγκαθιδρυθεί μια ευρωπαϊκή κεντρική κυβέρνηση από την πίσω πόρτα και η εθνική κυριαρχία να χάσει κάθε νόημα. Η κυριαρχία σημαίνει ευθύνη. Και όταν έχουμε κακή δημοσιονομική πολιτική, νομισματική πολιτική, θα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη μας. Όταν ε, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να ε, αναλαμβάνει τις ευθύνες του και να μην ζει εις βάρος των άλλων. Πιστεύω πως έχουμε πάρει τον ε, κακό δρόμο. Δίνω το λόγο τώρα στους υπόλοιπους εγγεγραμμένους ομιλητές. Ο κύριος Χόκμαρκ καταρχήν για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω πως είναι σημαντικό να μιλήσουμε για χρηστή διακυβέρνηση με την έννοια ότι φυσικά είναι σημαντικό να πιεστούμε όλοι ώστε να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες αλλά μην ξεχνάμε ότι η κύρια καλή διακυβέρνηση που έχουμε εμεί στα χέρια μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και Φυσικά υπάρχουν ε, μειονεκτήματα ε, ένα από τα μειονεκτήματα είναι το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Α μην το ξεχάσουμε πριν φτιάξουμε νέο νομοθεσίε ότι πρέπει να τηρήσουμε του πιο θεμελιώδει κανόνε. Αλλά να τονίσω και κάποια άλλα πράγματα που, αφορά τι χρηματοπιστωτικέ αγορέ. Α μιλήσουμε για τι χρηματαγορέ ω τμήμα τη οικονομία, όχι ω ένα ξεχωριστό τομέα. Γιατί ποτέ δεν θα έχουμε τι επενδύσει και νέε θέσει απασχόληση αν πιστεύουμε πω είναι χωριστή υπόθεση. Εγώ κάπως ενοχλήθηκα όταν διαπίστωσα ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής ε, Βασιλεία 2 θεώρησε πως οι νέοι κανόνες για τις κεφαλακές απαιτήσει θα μειώσει την οικονομική ανάπτυξη για 2, στο 2% και ότι αυτό είναι χαμηλό επίπεδο για εκείνον. Γιατί αν αυξάνουμε τις απαιτήσει τις κεφαλακές, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερες επενδύσεις και δεν το χρειαζόμαστε αυτό αυτή τη στιγμή αφού θέλουμε να δημιουργήσουμε νέα εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή οικονομία ενώ ταυτόχρονα θα βγούμε από τα δημοσιονομικά ελλείμματα που έχουμε. Και να τονίσω και κάτι που πραγματικά μπορούμε να κάνουμε από κοινού. Να δημιουργήσουμε δηλαδή την οικονομία της γνώσης. Είναι ένα παράδοξο ότι όσο περισσότερο οι κοινωνίες μας και οι οικονομίες μας τρέφονται προς την οικονομία της ε, γνώσης, τόσο λιγότερη εσωτερική αγορά έχουμε, γιατί αυτή διέπεται από κανόνες που αφορούν την βιομηχανία την παλαιού οικονομία, εκτό για τον τομέα των υπηρεσιών. Πρέπει να, συνεχίσουμε, έχουμε μια οδηγία για τις υπηρεσίες, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε μια μεταρρύθμιση που θα καταστήσει τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια πιο ανεξάρτητα, πιο ευρωπαϊκά, ανοιχτά για τους φοιτητέ και του ερευνητέ και να δημιουργηθεί μια δυναμική εξέλιξη στην κοινωνία τη γνώση. Α επιμένουμε σε όλα όσα μπορούμε να κάνουμε από κοινού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτή είναι η καλύτερη ε, ευρωπαϊκή διακυβέρνηση που μπορούμε να έχουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Χόκμαρκ. Η κυρία Λιούσκο έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ε, προέρχομαι από την ίδια χώρα με την σα, αλλά τίνω προς την αριστερά. Βλέπουμε την κατάσταση στην Ελλάδα, ε, γενική απεργία, ε, ε, διαμαρτυρίες στο, στους δρόμους, οργή για την όλη κατάσταση. Και αυτό έχει επιδεινωθεί επειδή ο, ο πυρήνα των χωρών του ευρώ έχουν ε, εγκαταλείψει την Ελλάδα. Αλλά η κρίση είναι μεταδοτική και μπορεί να ε, χτυπήσει και τις άλλες χώρες. Λίγες χώρες μπορούν να θεωρούνται ασφαλείς. Ε, θα πρέπει λοιπόν όλοι να ασχοληθούμε με την καταπολέμηση της κρίσης. Θα πρέπει να υποβάλουμε καλές προτάσεις, αλλά θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο που να σημαίνει ότι δεν ε, θα επιλέξουμε μόνο βράχοι πρόθεσμες λύσεις, ε, διότι έχουμε εδώ μια πυρκαγιά που καίει ό,τι βρει στον δρόμο της. Γι' αυτό θα πρέπει να ποντάρουμε σε λύσεις τέτοιες ώστε να διατηρηθεί η ζήτηση. Ε, και στόχο είναι πριν την διάσκεψη κορυφή του Ιουνίου να επιλεγεί η λύση που ανέφερε η προλαλή σα. Είναι σημαντικό η συνάντηση κορυφής ε, να να δώσει λύσεις ώστε να μην και με φλόγα οικονομίας η Ευρώπη θα πρέπει να διατηρηθεί η ζήτηση. Εγώ Απογοητεύτηκα πολύ με την μπλόφα περί ισότητας ε, που παρουσίασε ε, το τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών μετά την ε, συνεδρίασή του. Δεύτερον, θα πρέπει να θα πρέπει η κοινωνία μας να προσαρμοστεί στην αλλαγή του κλίματος. Θα πρέπει να αλλάξουμε δρόμο, θα πρέπει να αλλάξουμε κατεύθυνση. Είναι πολύ σημαντικό η Κομισιόν να δώσει στην κυρία Χέντεγκαρντ την ε, δυνατότητα να είναι πολιτικός για το κλίμα που να μπορέσει να επιφέρει πραγματικές αλλαγές. Τρίτον, όσον αφορά τις χρηματαγορές, ε, στην ε, Επιτροπή για την Κρίση είχαμε επίσκεψη από Αμερικανό καθηγητή πριν λίγο καιρό, ο οποίος είπε ότι δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τις χρηματαγορές διότι η Ευρώπη δεν το κάνει αυτό. Εκείνοι λένε δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τις ε, χρηματαγορές ε, ε, στη ΣΥΠΑ διότι δεν το κάνει και αυτό η Ευρώπη. Και η Ευρώπη λέει ότι δεν μπορεί να το ρυθμίσει επειδή ούτε και η ΕΠΑ κάνουν το ίδιο. Θα πρέπει λοιπόν να τολμήσουμε να επιφέρουμε τις αλλαγές αυτές. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κλίνς για 1,5 λεπτό. Κυρίες μου και κύριοι, στην πράξη μια στρατηγική είναι τόσο καλή όσο τα πραγματικά μέτρα που λαμβάνονται και οι ικανότητες εποπτείας και παρακολούθησης. Και εδώ μας οφείλει μια απάντηση η Κομισιόν. Θέλουμε στόχους με τους οποίους να μπορέσουμε να ταυτιστούμε. Αλλά θα πρέπει να είναι και συγκεκριμένοι. Μόνο αν είναι συγκεκριμένοι οι στόχοι αυτοί μπορούν να γίνουν δεκτοί και να επιτευχθούν. Ξέρω ότι στην αρχή των σκέψεων της Κομισιόν είναι η χρηματοπιστωτική κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει, η οποία έχει οξυνθεί με την κρίση στα, στα κρατικά οικονομικά. Είναι η πιο δύσκολη κρίση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Οι κρίσεις αυτές λοιπόν έχουν τροποποιήσει σημαντικά το σκηνικό. Αν λοιπόν μέσα στα επόμενα 10 χρόνια θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα, χρειαζόμαστε να έχουμε μια αλλαγή πορείας, να έχουμε ενιαία κριτήρια για να μπορέσει να επιτευχθεί αυτή η στρατηγική. Θα πρέπει να έχουμε ένα κοινό χρηματοοικονομικό πλαίσιο και ένα μηχανισμό επίλυση κρίσεων που θα μα επιτρέψει ότι στο μέλλον δεν θα ξαναβρεθούμε στην ίδια αυτή κατάσταση, αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε κατά κάποιο τρόπο μία πρόβλεψη καιρού για το μέλλον. Έχουμε την έκθεση Μάριο Μόντι σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών και εκεί παρουσιάζονται με πιστικό τρόπο οι, τα επιχειρήματά του ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μια, μια προσθήκη δημοσιονομικής πολιτικής στην κοινή νομισματική πολιτική. Και θα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν με ποιο τρόπο οι αποκλήσεις στον οικονομικό τομέα που έχουμε δει μέσα στα κράτη-μέλη θα αντικατασταθούν από μια πραγματική σύγκληση για να έχουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό εγχείρημα στον τομέα της οικονομίας και αυτό θα πρέπει να περιλάβει και τις μεταφορές και την ε, ενέργεια και τα συστήματα πλοήγησης. Είχατε 1,5 λεπτό μονάχα. Η κυρία Τούρουνεν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι οι εργασίε για τη στρατηγική 2020 είναι πολύ σημαντική διότι πρέπει να ε, συλλογιστούμε σοβαρά ε, από τι θα ζούμε στην Ευρώπη στο μέλλον και πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά τι θα κάνουν τα 23 εκατομμύρια άνεργων Ευρωπαίων στο μέλλον. Αλλά γενικά εμείς ως πράσινοι δεν έχουμε συγκεκριμένους στόχους σε σημαντικούς τομείς που θα κάνουν την κοινωνική Ευρώπη σε ε, ε, ε, προτεραιότητα τα επόμενα δέκα χρόνια. Καταρχήν θέλουμε να μειωθεί η ανεργία των νέων που σε όλα τα κράτη-μέλη είναι πολύ ψηλή. Θα πρέπει να εισάγουμε μια εγγύηση για τους νέους που θα ε, πρέπει να ε, εδραιώσει τη θέση των νέων στην ε, αγορά εργασία. Δεύτερον, θέλουμε συγκεκριμένου στόχου για την καταπολέμηση τη στόχια. Είναι ντροπή εάν τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην πιο πλούσια περιφέρεια του κόσμου δεν μπορούν να συμφωνήσουν για συγκεκριμένου στόχου για τη μείωση τη στόχια. Κάποιοι λένε ότι δεν του αρέσει ο ορισμό. Σε αυτού θα ήθελα να πω μην αφήσετε τα τεχνικά θέματα να είναι εμπόδια. Άλλοι λένε ότι δεν έχουμε τη νομική βάση στη συνθήκη. Έχουμε όμω νέα συνθήκη της Λισαβόνας. Τρίτον, θα πρέπει να εργαστούμε ε, με συνέπεια πάνω σε ένα ε, σχέδιο απασχόλησης. Θα πρέπει ε, να κατευθύνουμε πράσινε επενδύσει προ νέε θέσει απασχόληση και να ενθαρρύνουμε του νέου να ε, πάρουν τι θέσει απασχόληση αυτέ. Και τέλο, θα πρέπει ε, οι αρχηγοί κρατών να ε, θέσουν ως συγκεκριμένο στόχο μια κοινωνική Ευρώπη όπου η απασχόληση και η ασφάλεια θα είναι σημαντικά και θα πρέπει να φροντίσουμε όχι μόνο για την ποσότητα αλλά και για την ποιότητα των, των θέσεων απασχόληση. Αυτέ τι παραμέτρου θέλουμε να δούμε, αυτού του συγκεκριμένου στόχου παραμένει ακόμα δουλειά να γίνει. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, συνάδελφοι, να, ε, μείνετε, να παραμείνετε εντό του χρόνου ομιλία σα. Ο κύριο Χάρμπορ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να μιλήσω για την έλλειψη φιλοδοξίας που βλέπω στη στρατηγική για το 2020 τη Ευρωπαϊκή Ενώση. Για το πώς να χρησιμοποιήσουμε τα τωρινά μέσα, την ενιαία αγορά, να την κάνουμε να λειτουργήσει πράγματι αποτελεσματικά και να δημιουργήσουμε τις νέες θέσεις εργασίας και τις δυνατότητες αυτό που μίλησε, επανέφερε η προλαλήσασα. Δεν αρκεί και το λέω αυτό προς τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο, αν ακούει η Επίτροπος. Η ενιαία αγορά και τα επιτέγματά της να μπουν στο κεφάλαιο ε, κολλήματα και χαμένες διασυνδέσεις. Είναι πολύ πιο σημαντική η αγορά από αυτό και δεν αρκεί να λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει δράση. Είναι κοινή προσπάθεια των κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή μου, η Επιτροπή Εσωτερική Αγορά, ενέκρινε μια έκθεση αυτήν την εβδομάδα με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, η οποία στέλνει πραγματικά φιλόδοξε ιδέε για κοινέ δράσει για να ολοκληρωθεί η ενιαία αγορά. Θα τη λάβετε την επόμενη εβδομάδα με την έκθεση του καθηγητή Μόντι. Και α δούμε θεμελιώδει αλλαγέ να γίνουν και από τις δύο πλευρές. Αυτό που θέλουμε είναι μια ενία αγορά, μια πράξη για την ενία αγορά, δηλαδή σαφείς πολιτικούς ε, στόχους για την ολοκλήρωση της ενίας αγοράς και θέλουμε να δούμε και τις προμήθειες, τις δημόσιες προμήθειες. Ένα εργαλείο που το χρησιμοποιούμε ελάχιστα για να πετύχουμε την πράσινη τεχνολογία και την κοινοτομία, αυτού του στόχου. Δεν αναφέρεται σε αυτό το εγγραφό. Για όνομα του Θεού, γιατί μιλάμε για του άλλου στόχου όταν δεν κινούμεθα σε αυτά που ήδη έχουμε στα χέρια μα. Ευχαριστώ. Η κυρία Φιγκουερέιδο έχει το λόγο. Ενάμιση λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η στρατηγική δεν δίνει καμία απάντηση στα σοβαρά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Ακόμα λιγότερο στην πραγματική οικονομική και κοινωνική κατάρρευση που αντιμετωπίζουμε σήμερα σαν αποτελέσμα της πολιτικής ελευθερού ανταγωνισμού σε πολλά κράτη-μέλη, στις πιο εύθραυτες οικονομίες. Είναι λάθος να επιμένουμε σε ταυτόσιμες πολιτικές με την νεοφιλελεύθερη στρατηγική της Λισαβόνας. Δεν επετέθησαν οι στόχοι οι οποίοι αναφέρθηκαν της εξάλληψης της ένδυας και της πλήρους απασχόλησης. Όλα αυτά ήταν θύματα στο βωμό των κερδών των οικονομικών ομήλων σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Όλα αυτά ήταν τα αποτελέσματα της μηχανιστικής εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητος και της φιλελευθεροποίησης και της ιδιωτικοποίηση νευραλικών τομέων και δημοσίων υπηρεσιών για να υπάρξει ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών ομήλων στις ε, μεταφορές και στα ταχυδρομεία. Αυξήθηκε οι θέσει με μεγαλύτερο επισφαλή χαρακτήρα και η ανεργία η οποία αυτή τη στιγμή φτάνει τα 23 εκατομμύρια ε, ανέργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αποτέλεσμα υπάρχουν 85 εκατομμύρια άτομα σε κατάσταση ένδυας. Δείχνουν λοιπόν όλοι οι δείκτες ότι η συνέχιση αυτών των στρατηγικών που έχουν ακολουθεί μέχρι τώρα έχουν αποτέλεσμα χαμηλού ρυθμού αύξηση και χαμηλότερου ρυθμού ανάπτυξη από άλλε περιοχές του κόσμου, κατά το οποίο σημαίνει ότι θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο η ένδυα, η επισφαλής εργασία και ο κοινωνικός αποκλεισμό. Δυστυχώ, ο ευρωπαϊκός προπολογισμό δεν δίνει καμία απάντηση και δεν δημιουργεί την απαραίτητη οικονομική και κοινωνική συνοχή, όπως καταδεικνύει σαφώς η κατάσταση στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Είναι καιρό να καταλάβουμε λοιπόν τι συνέπειε αυτών των πολιτικών. Θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην κοινωνική βιωσιμότητα. Θα πρέπει να σταματήσει η κερδοσκοπία στο χρηματοοικονομικό τομέα και να ξαναγυρίσουμε στην πραγματική οικονομία. Θα πρέπει να σταματήσει να υπάρχει το σύμφωνο σταθερότητα και να ελέγξουμε τι ε, αλόγιστες ενέργειες του χρηματοπιστωτικού τομέα για να έχουμε κοινωνική ανάπτυξη. Next time I... Ευχαριστώ. Την άλλη φορά θα σας περικόψω, θα σας απο... αφαιρέσω το λόγο. Κύριος Μποργέζιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το γεγονός ότι είμαστε εδώ και συζητάμε και εξετάζουμε το περιεχόμενο της στρατηγικής για το 2020 ενώ στην Αθήνα ε, σε ένας λαός ολόκληρος οι εργάτες είναι στα όρια του γκρεμού αυτό προσφέρει μια εικόνα αρκετά σημαντική θα τολμούσα να έλεγα χονδροειδή ε, εικόνα όσον αφορά την πολιτική της Ευρώπης. Είναι μοναδικό σε μετρήτη κατάσταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην αισθάνεται το καθήκον να προβεί σε ενδελεχή προβληματισμό και αυτοκριτική. Δεν είναι ότι δεν βλέπει ότι αυτή η κατάσταση της κρίσεως, αυτή η κατάσταση που αποκτά χαρακτήρα δραματικό από κάποιες στοιχές, είναι συνέπεια πολλών και σοβαρών σφαλμάτων, όπως αποδεικνύει και η χροκοπία της στρατηγικής της Λισαβόνας. Πολλά λάθη, πολλά σφάλματα και υπάρχει και ένας ένοχος που είναι το ευρώ. Σε όλες τις δηλώσεις λέγεται ότι είναι μεμονωμένη η Ελλάδα. Ελπίζω να μην γίνει, αλλά ίσως να συμβεί το ίδιο και στην Ισπανία και αυτό θα είναι μεμονωμένη υπόθεση. Εδώ ακολουθούμε και μεμονωμένες δικαιολογίες και είναι μεμονωμένα και τα subprime. Είναι λίγο, ελάχιστα αξιόπιστο, δύσκολο να αποδεχτεί κανείς τις αναφορές Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποφάσισε να καθαρίσει, να ξεκαθαρίσει τις ευρωπαϊκές τράπεζες και να πείσω από ταμιευτές, τους παραγωγούς, στην πραγματική οικονομία τι βρωμιά υπάρχει ακόμα εντό των ευρωπαϊκών τραπεζών για να διαμορφωθεί μια στρατηγική. Πρέπει να έχουμε υπόψη αυτά τα σημεία να τα θυμηθούμε και πρέπει να θυμόμαστε ότι μια στατική σοβαρή πρέπει να ξεκινεί από την πραγματική οικονομία, από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα πρέπει να δώσει ένα ρόλο μέσω της συμμετοχής υπευθυνότητα μέσω συμμετοχής των εργατών, των εργαζομένων. Ευχαριστώ ο κύριος Σιέγκεντη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η τωρινή κατάσταση δεν είναι κάτι το οποίο, για το οποίο φταίνε ούτε οι εργαζόμενοι ούτε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο υπεύθυνο είναι η φιλοσοφία που έχει ακολουθηθεί μέχρι τώρα στον οικονομικό τομέα που έχει θέσει στο κέντρο της τους μεγάλους χρηματοοικονομικούς ομίλους και τις μικρές χώρες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τις έχει θέσει στο περιθώριο. Οι πολυεθνικές εταιρείε θέλουν να δημιουργήσουν το μεγαλύτερο δυνατό περιθώριο κέρδους για τον εαυτό τους, τον ευρύτερο δυνατό χώρο δράσης για τον εαυτό τους, ώστε να αυξήσουν και την κερδοφορία τους. Η στατηγική μας αντίθετα θα πρέπει να εστιάσει στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και το κόμμα μας, το Γιόμπιξ στην Ουγγαρία, θέλει να σπάσει η επικυριαρχία των μεγάλων επιχειρήσεων και των μεγάλων ομίλων. Πρέπει να έχουμε την Ευρώπη των οικογενειών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μια Ευρώπη η οποία είναι κοντά στον απλό πολίτη. Ευχαριστώ πολύ και ο Ρόιλ έχει το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Προεδρία και ο Πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι δεν μπορούμε να λειτουργούμε το σύνθημα σώζον αυτό σωθήτο». Ε, χρειαζόμαστε ένα ε, γενικό σχέδιο και γι' αυτό χρειαζόμαστε και στρατηγική για τη δράση. Ωστόσο, με το πρόγραμμα αυτό το 2020 και όσον αφορά τον τρόπο πώς θα καταλήξουμε σε αποτελέσματα, κατά τη γνώμη μου δεν πρόκειται για στρατηγική. Είναι συλλογισμοί που έγραψε κάποιο σε χαρτί και που θα θέλουμε να υιοθετήσουμε με μια γρήγορη διαδικασία. Ο πρόεδρο τη Επιτροπή είπε κάτι πολύ σωστό. Είπε ότι το πρόβλημα με την στρατηγική τη Λισαβόνα είναι ότι οι συμμετέχοντε δεν ένιωσαν ότι είναι δικοί του, δεν συμμετείχαν κατά την εκπόνησή τη και γι' αυτό δεν πέτυχε. Και πράγματι έτσι έχουν τα πράγματα. Εάν όμω συμβαίνει αυτό, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο που απαιτεί ε, να συμμετάσχουν οι συμμετέχοντες, οι ενδιαφερόμενοι, να συζητήσουμε επαρκώς ώστε να έχουμε μια καλή στρατηγική. Η κριτική που ακούγεται είναι ότι ε, ε, αφήνουμε να μας υπαγορεύσουν εδώ στο Κοινοβούλιο τι πρέπει να κάνουμε. Επανειλημμένα έχει εκφραστεί η επιθυμία ε, το πρόγραμμα να εκπονείται ε, πιο προσεκτικά. Αλλά ε, αντί για αυτό η διαδικασία συνεχώς συντομεύεται. Το συστάμε σήμερα, το συστήσει το Συμβούλιο τον Ιούνιο και πάει τελείωσε. Μη σας κάνει εντύπωση αν τελικά δεν υπάρξουν αλλαγές στο εμπόριο. Δεν μπορεί να επιφέρει κανείς έτσι αλλαγές. Χρειάζεται μια εντελεχής ανάλυση και όχι κάποιες ε, επιφανειακέ ε, συνέπειε, ε, όπως κάνει η Επίτροπος για το κλίμα αυτές τις μέρες. Ε, θεωρεί δηλαδή ότι μπορούμε πολύ εύκολα να πετύχουμε το στόχο του 30-40% όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε προσεκτικά την κατάσταση και μετά να δούμε προσεκτικά τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε όσον αφορά την καινοτομία, την οικονομία, ε, την έρευνα κλπ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σέρκας, δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Λόπες Καρίδο και ευχαριστώ και την Επιτροπή. Ελπίζω ότι θα υπάρξει κάποια συνέχεια στα λόγια σας και το Συμβούλιο του Ιουνίου θα είναι πολύ διαφορετικό από το Εαρινό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, γιατί αυτά τα οποία αναφέρετε δεν με καταπραίνουν, δεν μου δίνουν τη δυνατότητα να φανταστώ ένα Συμβούλιο το οποίο δεν θα είναι γεμάτο από αμφιβολίες και το οποίο θα αμφιταλαντεύεται. Θέλουμε να έχουμε πολιτικούς στόχους οι οποίοι να είναι όχι απλώς βολικοί αλλά πρέπει να είναι εφικτή. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Λόπε Γκαρίδο και σα ευχαριστώ για την βοήθεια που έδωσε η Ισπανική Προεδρία για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα θέματα. Έχουμε ιστορικέ στιγμέ που διατρέχουμε στην ιστορία τη Ευρώπη. Έχουμε μεγάλε προκλήσει να αντιμετωπίσουμε στην επόμενη δεκαετία. Θέλουμε περισσότερη Ευρώπη ή λιγότερη Ευρώπη. Αυτό είναι ο στόχο τη στρατηγική 2020. Είτε θα είμαστε πιο ενωμένοι σε 10 χρόνια, είτε θα είμαστε λιγότερο. Για να είμαστε πιο ενωμένοι όμως θα πρέπει να από κοινού να αντιμετωπίσουμε τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, αλλιώς θα επανέλθουμε νομοτελειακά στην εποχή των εθνικισμών και θα χάσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα. Ας είμαστε λοιπόν αλληλέγγυοι, ας ακολουθήσουμε το στόχο της αλληλεγγύης και της πιο ισοδίκαιας κατανομής του πλούτου που θα δημιουργηθεί, αλλιώς θα τα αφήσουμε <clears throat> όλα στα χέρια των αγορών. Εγώ δεν νομίζω ότι όλα αυτά έγιναν επειδή υπήρχε υπερβολική ρύθμιση, υπερβολική κοινωνική δικαιοσύνη στην Ευρώπη. Κάθε άλλο. Η έλλειψη κοινωνική δικαιοσύνη, η έλλειψη ρύθμιση ήταν αυτή που οδήγησε στην κρίση. Κρατήστε του στόχου σα για μία αντιμετώπιση τη ένδυα, για περισσότερη εκπαίδευση και κατάρτιση που βρίσκεται στο κείμενο τη Κομισιόν, αλλά όχι του Συμβουλίου, και α συμμετέχει και το Κοινοβούλιο σε όλα αυτά, ώστε να ακούγεται και η φωνή των πολιτών και όχι μονάχα η φωνή των ηγετών ή των <clears throat> λεγόμενων αγορών που πολλές φορές είναι απλώς μια φενάκι για τους κερδοσκόπους. Ευχαριστώ κύριο Σιμετή, μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι πρόβλημα όλων μας και των χωρών που δεν συμμετέχουν στο ευρώ. Η Ευρώπη σήμερα ε, χρειάζεται συντονισμένη και ισχυρή δράση, όχι ε, περαιτέρω κατακαιρματισμό. Γι' αυτό είναι δυσάρεστο ότι 11 χώρες δεν θα συμμετέχουν την Παρασκευή. Η Ευρώπη έχει κοινή μοίρα, αλλά αυτό δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή. Η εποπτεία των χρηματαγορών θα πρέπει να ενισχυθεί. Θα πρέπει να εφαρμοστεί πιο αυστηρή νομοθεσία. Και εγώ ως φιλελεύθερος το βλέπω αυτό και το παραδέχομαι. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει με ισορροπημένο τρόπο. Θα πρέπει να υπάρξει διεθνής συντονισμό. Να ενεργήσουμε ε, ισχυρά και επιθετικά, αν είναι απαραίτητο, αλλά όχι σε πανικό. Θα πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι όσο γίνεται, για να μην βλάψουμε περαιτέρω την οικονομική ανάπτυξη που παρόλα τα προβλήματα, παρά το πρόβλημα της Ελλάδας, ε, πιστεύω ότι θα μπορέσει να βελτιωθεί. Κύριε Πρόεδρε, όταν άκουσα τον ε, κύριο Μπλουμ, ταράχτηκα, δεν βρίσκεται εδώ σήμερα, αλλά η σύγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Σοβιετική Ένωση είναι προσβολή όλων όσων υπέφεραν ε, υπό Σοβιετική τυραννία και αυτών που πέθαναν. Ε, πιστεύω ότι ο κύριος Πλούμ θα πρέπει να ε, ζητήσει συγγνώμη να απολογηθεί απέναντι στους ανθρώπους που προσέβαλε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Ο κύριος Μπόκρος είναι επόμενος για ένα λεπτό όταν ο Ισπανός Πρωθυπουργό Χωσέ Λουίς Ροδρίγες Σαπατέρο εγγενίασε την Ισπανική Προεδρία στην, στο Στρασβούργο έκανε μια ομιλία και αναφέρθηκε στην Ευρώπη για το 2020. Δεν ανέφερε, δεν είπε λέξη γιατί στο καλό πέτυχε εν πρώτη στρατηγική της Λισαβόνας και το έθεσα το ερώτημα πώς μπορεί κανείς να αναλύσει και να καταλήξει σε νέα στρατηγική χωρίς να αναλύσει το που απέτυχε η προηγούμενη στατηγική. Δεν έχω επιλογή παρά να επαναλάβω το ερώτημά μου. Διότι το νό έγγραφο κουβέντα δεν λέει περί της αποτυχίας και περί των λόγων της αποτυχίας. Λοιπόν, παρακαλώ κύριε Γαρίγα, αν μπορείτε απαντήστε το ερώτημά μου. Γιατί είναι δυνατόν και πώς είναι δυνατόν να δημιουργήσει κανείς πολύ φιλόδοξους νέους στόχους χωρίς να αναλύσει, να αναλύσει πριν για ποιους λόγους απέτυχε η στρατηγική της Λισαβόνας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μπόκρος. Ο κύριος Ντεγιόγκ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Πρόεδρε, πιστεύω ότι η Κομισιόν και το Συμβούλιο έχουν λάβει σαφείς αποφάσεις όσον αφορά ε, την ε, δημοκρατία. Θα ήθελα πολύ να ξέρω πώς αποφασίζει η, το Συμβούλιο. Η νομοθεσία στα κράτη-μέλη εδώ και ε, δέκα χρόνια πραγματοποιείται με τρόπο ε, όπου δεν ε, συμμετέχουν οι πολίτες ταυτόχρονα. Λέμε ότι θέλουμε μεγαλύτερη ποσόστοση για την απασχόληση, αυτό θα ήταν πολύ ωραίο, αλλά δεν θέλουμε να υπάρχουν ακόμα περισσότεροι φτωχοί εργαζόμενοι. Και όσον αφορά τις ε, δημόσιες δαπάνες. Πώς μπορούμε να εγκρίνουμε προϋπολογισμό που να αυξάνεται μόνο κατά 5,8% όσον αφορά, ε, κατά αφορά την ε, κοινωνική εσωτερική αγορά. Πώς μπορούμε να κάνουμε πιο κοινωνική την εσωτερική αγορά Μπορούμε να το κάνουμε αυτό με τις ε, δημόσιες προμήθειες και τα δημόσια ε, έργα. Και όσον αφορά την ε, καταπολέμηση της φτώχειας, αυτό θα γίνει με την ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά αυτή συνήθως έχει σαν αποτέλεσμα οι διευθυντές να παίρνουν περισσότερα χρήματα, όχι όμως οι εργαζόμενοι. Ευχαριστώ. Η κυρία Βιτσότο, για να λύσουμε το πρόβλημα τη απασχόληση επικοδομητικά, θα έχουμε τρει λέξει να χρησιμοποιήσουμε. Να αντιδράσουμε, να εξελιχθούμε και να προστατεύσουμε. Να αλλάξουμε ε, την Ευρωπαπαγάνδα να αντιμετωπίσουμε με συγκεκριμένο τρόπο τα προβλήματα που πλήττουν του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, με στι διάσταση μεταξύ του τρόμου, τη κατάρ... του κόσμου της κατάρτισης και των αναγκών της αγοράς και να δώσουν τους νέους ε, να αλλάξουν άποψη για τις χειρονακτικές εργασίες. Θέλουμε μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020 που να είναι κάτι θετικό και να ε, συμβάλλουν και, και εργαζόμενοι και επιχειρήσεις. Να, θα πρέπει να υπάρξει σταθερότητα στον αφορά τις θέσεις απασχόλησης. Προστασία. Σε, να δώσουμε δουλειά σε αυτούς που την έχασε, κυρίως πολίτες θα πρέπει τα κάτι μέλη να αξιολογήσουν τι πολιτικέ τη μεταναστευτικέ βάσει των πραγματικών αναγκών τη μετανάστευση. Έχουμε 3 εκατομμύρια ανέργους, 23 ε, εκατομμύρια ανέργους. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε κατά πόσο θα πρέπει να εργάζονται οι εξοκοινοτικοί. Και θα πρέπει να εξετάσουμε και το κοινωνικό μας σύστημα. Χρειάζεται θάρρος, αποκέντρωση και νέα μέτρα θαραλέα. Ευχαριστώ. Κύριος Μαρινέσκο έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη απαιτεί επενδύσεις οι οποίες είναι μαζικές και συνεκτικές μεταξύ άλλων και στον τομέα των μεταφορών που είναι το 6% του ΑΕΠ όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίνουν εργασία σε πάνω από 10 εκατομμύρια ανθρώπους η Κομισιόν και το Συμβουλίο στην προετοιμασία του εγγράφου του για τη στρατηγική του 2020 θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα εξή στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά στο τομέα των μεταφορών. Πρώτα απ' όλα, να προωθήσουμε τι επενδύσει και την ανάπτυξη για να μπορέσουμε να επιτύχουν την πράσινη, τις πράσινες μεταφορές, να βοηθήσουν να μειωθούν οι εκπομπές άνθρακος, διοξιδίου του άνθρακος με την λεγόμενη ETS, την ευφυά διαχείριση των μεταφορών, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τη διαχείριση των τη εναέρεια κυκλοφορία. Επίση, να υπάρξουν κατάλληλε υποδομέ για να προστατευτεί το περιβάλλον, οι εργαζόμενοι και φυσικά και η ασφάλεια των επιβατών. Και ένα ιδιαίτερο τομέα που θέλω να υπογραμμίσω αφορά τα εξή στοιχεία που μου φαίνονται πάρα πολύ σημαντικά. Να υπάρξει η εφαρμογή των ανοιχτών και ενιαίων ουρανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η επίτευξη τη διαλειτουργικότητα στον τομέα των σιδηροδρόμων, η ασφάλεια στις οδικές μεταφορές, η εφαρμογή της καλής διαχείρισης των εσωτερικών υδάτινων δρόμων και λιμένων, η αυτοκινητόδρομη της θάλασσας και η βιώσιμη ανάπτυξη στον τομέα της αστικής κινητικότητας. Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των μεταφορών και της κινητικότητας. Θα πρέπει να αποτελέσουν λοιπόν το κομβικό τμήμα της στρατηγικής 2020 για να έχουμε μία ανάπτυξη συντονισμένη και βιώσιμη στον τομέα των μεταφορών και δημιουργία θέσεων εργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Ποδηματά για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα ως Ελληνίδα να εκφράσω τη βαθιά μου λύπη για τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν σήμερα στη χώρα μου με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις πολίτες που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε μια τράπεζα όταν ακραία στοιχεία που παρισύφρισαν σε μια μεγάλη αλλά απολύτως ειρηνική διαδήλωση έβαλαν φωτιά. θέλω λοιπόν με αυτή την ε, τραγική αφορμή και επειδή γνωρίζω ότι όλη η ευρώπη και όλα τα ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης παρακολουθούν σήμερα την ελλάδα να ζητήσω από όλους εδώ από όλους τους συναδέλφους υπευθυνότητα σοβαρότητα αλληλεγγύη και κυρίως σεβασμό απέναντι σε ένα λαό που περνάει πολύ δύσκολες στιγμές. και τα λέω αυτά αγαπητοί συνάδελφοι διότι φοβούμαι ότι από αύριο θα σπεύσουν ορισμένοι σε μεγάλες ευρωπαϊκές εφημερίδες σε ορισμένες πρωτεύουσες να υποστηρίξουν με αφορμή ακριβώς αυτά τα τραγικά γεγονότα ότι δικαιώνονται οι φόβοι και οι αμφιβολίες τους για το αν η ελλάδα είναι αποφασισμένη και μπορεί να φέρει σε πέρας τις πολύ δύσκολες αποφάσεις που έλαβε για τη δημοσιονομική προσαρμογή γιατί ήδη από την επόμενη μέρα τη συμφωνία τη περασμένη Κυριακή άρχισε πάλι η ίδια ιστορία που την παρακολουθούμε από τις 11 φεβρουαρίου και μετά με σειρά σχολείων για την αναποτελεσματικότητα των ελληνικών μέτρων για την προοπτική αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέου με το ενδεχόμενο ακόμα και εξόδου της χώρας από τη ζώνη του ευρώ και βεβαίως με νέες επιθέσεις από τις αγορές σε βάρος όχι μόνο των ελληνικών ομολόγων αλλά και των πορτογαλικών και των ισπανικών. και διερωτώ με αγαπητοί συνάδελφοι μια που συζητάμε και για την προοπτική της στρατηγικής του 2020 πού θα πάει αυτό πού θα πάει δηλαδή αυτή η απόλυτη εξάρτηση εθνικών οικονομιών από τις κρίσεις των αγορών από τις αξιολογήσεις οίκων πιστοληπτικής ικανότητας που δεν λογοδοτούν πιθανά, δεν υφίστανται απολύτως καμία συνέπεια και έλεγχο για τις αξιολογήσεις τους είτε είναι σωστές είτε λάθος είτε αφορούν επιχειρήσεις είτε κράτη και μάλιστα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ. ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Μανέσκου. Ένα μισή λεπτό ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε αντιμετωπίσει μια κρίση που είναι η πιο σοβαρή της ιστορίας της παγκόσμιας οικονομίας. Είναι απαραίτητο οι προσπάθειές μας να κατευθυνθούν καλύτερα για να δώσουμε μια αύξηση παραγωγικότητας και ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και εν τέλει την οικονομική ανάπτυξη. Οι στόχοι του 2020 για να είναι ρεαλιστικοί θα πρέπει να καθοριστούν σε συνέργεια με τους στόχους που έχουν θέσει τα κράτη-μέλη επί τη βάση των δικών τους προτεραιοτήτων και ιδιαιτεροτήτων. Γι' αυτό θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να διαμορφώνονται και να ακολουθούν τους εθνικούς στόχους η Κομισιόν θα πρέπει να παρουσιάσει νέα μέτρα και ενδεχομένως και κυρώσεις για αυτούς που δεν εφαρμόζουν τη νέα στρατηγική και περαιτέρω κίνητρα για αυτούς που την χρησιμοποιούν τη στρατηγική αυτή. Τα μέτρα αυτά λοιπόν θα πρέπει να ακολουθούν τους στόχους οι οποίοι έχουν θεσπιστεί και φυσικά να πριτανεύει η αρχή της τη συμβατότητα με του εθνικού στόχου. Θα πρέπει φυσικά να έχουμε και πολιτικέ συνοχή για να επιτευχθούν οι οικονομικοί και κοινωνικοί στόχοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ προσεκτικά τι προτάσει Κομισιόν, παραδείγματο χάρη την αμέση αναστολή τη παροχή διαφορετικών ταμείων, εάν τα κράτη-μέλη έχουν υπερβολικό έλλειμμα του προπολογισμού. Εδώ θεωρώ ότι ένα τέτοιο μέτρο όμω είναι τελείω αντίθετο με το στόχο τη συνοχή που είναι να μειωθούν ακριβώ οι αποκλήσει μεταξύ 100 μελών. Ευχαριστώ, λέω ε, κύριος Βλασάκη, ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το πληθυσμό είναι η μεγαλύτερη γεωπολιτική οντότητα στον κόσμο. Οι οικονομίες μας έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσονται με βάση την καινοτομία και τις εξαγωγές. Θα πρέπει όμως ε, να ε, είμαστε μετριόχρονες απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ε, την Ιαπωνία, την Ινδία και την Βραζίλια. Πιστεύω ότι η στρατηγική μας θα πρέπει να συνεχίσει να επικεντρώνεται στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Τα κοινωνικά θέματα και η αλλαγή του κλίματος δεν θα πρέπει να αποσπάσει την προσοχή μας από τους βασικούς αυτούς στόχους. Ταυτόχρονα χρειαζόμαστε Χρειάζεται να καταλάβουμε ότι η ε, ευφυή ανάπτυξη στην, ε, στα κράτη-μέλη, στι περιφέρειες ε, και στι τοπικέ κοινωνίε, δεν είναι δυνατή χωρίς την απαραίτητη υποδομή, την υποδομή μεταφορών, την περιβαλλοντική υποδομή. Η στρατηγική 2020 δεν καλύπτει ικανοποιητικά τους τομείς αυτούς, ούτε καλύπτει ικανοποιητικά την ανάγκη για συνεχείς επενδύσεις στις υποδομές στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες που δεν έχουν αναπτυχθεί αρκετά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Higgins για ένα λεπτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ετοιμάσει στρατηγική μέχρι το 2020 και βασίζεται σε ενοφιλελεύθερο καπιταλισμό και στο σύστημα της αγοράς. Με άλλα λόγια, στους ίδιους παράγοντες που βήθησαν τον κόσμο στην παρούσα οικονομική κρίση, στο χάος και η ανταπόκριση των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκή Ενώση αφορά την χρηματοπιστωτική κρίση στην Ελλάδα έδειξε ότι υπεχώρησαν στου κερδοσκόπου και, και στι καρχαρίε του χρηματιστηριακού κόσμου. Ε, θα πρέπει οι συνταξιούχοι και οι φτωχοί της Ελλάδας να περικόψουν τα εισοδήματά τους για να τροφοδοτήσουν ε, τη λεμαργία αυτών των χρηματιστικών αγορών που δεν είναι ένας θεός όπως τον παρουσιάζουν τα μέσα ενημέρωσης αλλά επενδυτικές τράπεζες, ε, μέτοχοι κλπ. Παράσιτα που θέλουν υπερβολικά τεράστια κέρδη κερδοσκοπώντας κόπημα για να δημιουργήσουν χρηματοπιστωτική αστάθεια και να εκμεταλλευτούν αυτή και να ροφήξουν το αίμα των εργαζομένων. Αυτή την Ευρώπη θέλουμε για το 2020. Είναι παθητικά αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Μπαρόσο. Γιατί αυτά που ακούσαμε να ζητάει υπευθυνότητα. Είναι να σαν ζητά τον Καρχαρία να σταματήσει να θέλει πιει αίμα. Θα πρέπει να υποστηρίξουν όλοι οι εργάτε στην Ευρώπη τη μάχη του ελληνικού εργατικού κινήματο. Ε, δεν πρέπει βέβαια οι ηλίθιοι να κάψουν τράπεζε για να δράσει το σύστημα. Χρειάζεται όμω σταθερή κινητοποίηση, να κινητοποιηθούν, να στηριοποιηθούν οι εργαζόμενοι και αυτό το άλλο στο σύστημα να αντικατασταθεί με δημοκρατικό σοσιαλισμό και μια πραγματική ανθρώπινη κοινωνία που θα πρέπει να δημιουργηθεί μέχρι το 2020. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πάσκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με κάθε σεβασμό προς τα έγγραφα που έχουμε στη διάθεσή μας είναι πολύ δύσκολο να παραγνωρίσουμε την ομοιότητα που παρουσιάζουμε με ορισμένα σχέδια πενταετούς χαρακτήρα σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. θεωρούσαν ότι ήταν αξιόπιστα και προσπαθούσαν να πείσουν το λαό ότι θα λειτουργήσουν. Αλλά κάθε φορά απετύχανε στρατηγική και καταβυθιζόταν η οικονομία διότι δεν σεβαζόταν τους βασικούς κανόνες της οικονομικής επιστήμης. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή αγωνίζεται τη στιγμή που έναντι της Κίνας και της Ινδίας έχει ένα πιο μορφωμένο πληθυσμό και ο βασικός λόγος γι' αυτό είναι το γεγονός <clears throat> ότι το Ευρωπαϊκό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο τους αρέσει να δημιουργούν νέα θεσμικά όργανα, νέα γραφεία. Εκατομμύρια μορφωμένων ανθρώπων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε καινοτόμους και ε, δημιουργικούς τομείς περνάνε τον καιρό τους πρόχνοντας χαρτιά σε δημόσια και άλλα γραφεία και καταδαπανώντας δημόσια χρήματα. Αν θέλουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί θα πρέπει να απλοποιήσουμε τους κανόνες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο πνεύμα για το επιχειρήν, να μειώσουμε το άχθος που φέρνουν οι επιχειρήσει. να αφήσουμε περιθώριο για τη δημιουργικότητα των επιχειρηματιών και για την πρωτοβουλία. Ο κύριος Καράς. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η κοινή Ευρώπη, μια αξιόπιστη πολιτική ένωση, βιώσιμη απασχόληση, ε, η κοινωνική συνοχή και η βιώσιμη ανταγωνιστικότητα. Όλα αυτά είναι στόχοι μας. Η Ευρώπη 2020 δεν είναι ο στόχος μας. Η Ευρώπη 2020 είναι μέσο για να πετύχουμε τους στόχους. Έχουμε την, ε, θα πρέπει να γίνει η διακήρυξη Σούμαν μας για το έτος 2010 και θα πρέπει να είναι εξίσου συγκεκριμένη με τη δήλωση του 1950. Ε, δεν θα πρέπει να είναι ένας κατάλογος από επιθυμίες για το μέλλον που δεν μπορούν να εκπληρωθούν και να πνιγεί στα προβλήματα. Η Ευρώπη 2020 θα πρέπει να είναι ένα συγκεκριμένο μέσο το οποίο να ε, έχει επαρκή χρηματοδότηση και να αποτελέσει επαρκή ε, ανταπόκριση στην κρίση. Η Ευρώπη του 2020 θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένα προγράμματα για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την έρευνα, ε, την βιώσιμη ανάπτυξη. σε όλα τα κράτη-μέλη και η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βάλουμε το χέρι στο ταμείο για να έχουμε μια συγκεκριμένη βάση και θα πρέπει να ξέρουμε τι θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε και γιατί χρειαζόμαστε τα χρήματα. Χρειαζόμαστε επίσης στη στρατηγική, ε, στη στρατηγική Στη, στη, στην ε, Ευρώπη 2020 χρειάζεται να γίνει έλεγχος ε, ε σκοπιμότητας. Χρειαζόμαστε πλήρη υποστήριξη των μέτρων του Όλη Η Ευρώπη 2020 θα πρέπει να αποτελέσει έκφραση της νέας πολιτικής βούλησης και θα πρέπει να είναι η απάντησή μας ε, στον ε, αυξανόμενο εθνικισμό και προτεξιονισμό. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την εσωτερική αγορά και εκτός από την νομισματική ένωση να έχουμε και μια οικονομική ένωση που να αποτελούν μέρος μιας αξιόπιστης πολιτικής ένωσης. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε, τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κοφεράτη, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε ομολογώ την ανησυχία μου σχετικά με τη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου. Διότι στη συζήτηση δεν βλέπω στοιχεία καινοτομία που θα μπορούσαν να διορθώσουν τι συστάσεις της Ερηνής Συνόδου Κορυφή. Αυτές οι στάσεις ήδη ήταν απογοητευτικέ. Απογοητευτικέ δεν είχαν καμία σχέση με ένα ελάχιστο κριτικής αναλύσεως όσον αφορά τα όρια της Λισαβόνα, τι συνέπειε της έλλειψη εφαρμογής κάποιων σημαντικών πτυχών σε επίπεδο πολιτικό και πολιτισμικό. Απογοητευτικές, διότι ήταν απόμακρες από την κρίση. Ήταν κάποια σημεία γενικόλογα χωρίς να συνδέονται λογικά. Σύνολο άθροισμα καλών προθέσεων που δεν μπορούν να παραγάγουν πολιτική. Και εδώ ε, βρισκόμαστε ακόμα και δεν βλέπω συγκεκριμένη βούληση επιλογής προτεραιοτήτων. Το πρόβλημα της Ευρώπης είναι το επίπεδο ανταγωνιστικότητά της, ανταγωνιστικότητάς της στο παγκόσμιο ε, επίπεδο. Δεν μπορούμε να αποχωριστούμε από την κοινωνική συνοχή που είναι θεμελιώδης παράγοντας ανταγωνιστικότητας. Χωρίς συνοχή καμία χώρα και ακόμα λιγότερο τα υπερεθνικά σύνολα δεν μπορούν να σταθούν στην παγκόσμια αγορά διότι εντός θα υπήρχαν συγκρούσεις που θα οδηγούσαν στην απώλεια ανταγωνιστικών θέσεων καθημερινά. Και από την άλλη πλευρά είναι και το θέμα τη καινοτομία. Δεν αρκεί να αναφέρεται. Θα πρέπει να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι που δεν περιέχονται εδώ και δεν υπάρχουν εκεί πόροι που διατίθενται, θα πραγματευτούν για την καινοτομία και για το προϊόν και για τη διαδικασία. Μόνο η ποιότητα στη δουλειά, στην καθημερινή ζωή και στην παραγωγή των αγαθών και υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει την Ευρώπη σε θέση τέτοια που να μπορεί να ανταγωνιστεί μετά από τις σοβαρότητες συνέπειες αυτής της κρίσεως. Να προσθέσω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που δεν αναφέρθηκε ποτέ. Στόχοι φιλόδοξοι ε, μπορούν να υλοποιηθούν αν υπάρχει και πολιτική ολοκλήρωση. Δεν μιλάνε για αυτό τα κράτη-μέλη. Το ανέβαλα το θέμα. Η, χειρότερη, η χείριστη αυτή διαχείριση της ελληνικής κρίσεως απέδειξε την έλλειψη προσέγγιση αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Στρίτσεκ, ο κ. Στρίτσεκ, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε. Προέρχομαι από κράτος μέλος όπου μέχρι την ηλικία των 28-29 ετών ζούσα σε ένα σύστημα που βασιζόταν στον κεντρικό ε, προγραμματισμό. Η ζωή ε, πραγματοποιόταν με βάση πενταετή προγράμματα ε, και το ένα ακολουθούσε το άλλο, διότι κανένα τελικά δεν πέτυχε. Συγγνώμη που είμαι κάπω ευαίσθητο για τα θέματα του κεντρικού προγραμματισμού και σχετικά με την ιδέα του να ζωγραφίσουμε μια εικόνα της Ευρώπης το 2020. Ναι, είναι ενδιαφέρον αυτό, αλλά ε, μα τυφλώνει σε σχέση. Ε, δεν βλέπουμε αυτά που πραγματοποιούνται σήμερα και στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη. Ε, παρακολούθησα πολύ ε, στενά την συζήτηση εδώ στο Κοινοβούλιο. Ακούμε περισσότερη κεντρική διαχείριση, ε, κεντρικό προγραμματισμό. Και τη συγκεκριμένη στιγμή πιστεύω ότι χρειαζόμαστε λιγότερη συγκέντρωση, περισσότερη εμπιστοσύνη στην αγορά. Χρειαζόμαστε περισσότερη ελεύθερη αγορά. Χρειαζόμαστε μηχανισμού τη αγορά, διότι όλα όσα γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη και πέρα από αυτήν, στι Ηνωμένε Πολιτείε και αλλού, όλα αυτά αποτελούν παράδειγμα της αποτυχίας της κρατικής παρέμβασης. Ευχαριστώ. Δύο, Κυρία Δεκαστή Βέρα, δύο λεπτά ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολλοί από τους συναδέλφους οι οποίοι προελάλησαν θέτουν το ερώτημα του γιατί απέτυχε η ατζέντα της Λισαβόνας και μήπως θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την ανάλυση μιας τέτοιας αποτυχίας για να δούμε ποια πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα. Κατά τη δική μου άποψη το πρόβλημα της ατζέντα της Λισαβόνας είναι ότι τελικά ήταν μονάχα μια, ένα όραμα μέσα σε μια φυσαλίδα Δεν υπήρξε καμία πρακτική εξέλιξη αυτή τη ιδέα και τελικά καταλήξαμε στο να υπάρχει μια θεωρητική ενατένιση η ατζέντα της Λισαβόνας για την οποία όλοι, στην οποία όλοι αναφερόμαστε και συγχρόνως μια πρακτική η οποία δεν είχε καμία σχέση. Η στρατηγική λοιπόν 20-20 με την συσσωρευμένη εμπειρία από την αποτυχία της Λισαβόνας θα πρέπει να είναι μια νέα ατζέντα η οποία θα μπορέσει να προχωρήσει μονάχα αν υπάρχει μια πραγματική και στεναρή δέσμευση από την πλευρά όλων των θεσμικών οργάνων, πολιτικών θεσμικών οργάνων και των εθνικών πολιτικών οργάνων. Αν υπάρξει λοιπόν μια τέτοια δέσμευση <clears throat> θα πρέπει περαιτέρω να είναι μια δέσμευση επαληθεύσιμη η οποία θα μπορεί να επιβεβαιώνεται μέσω της κοινή πορείας και της δυνατότητος τροποποίησης πορείας όταν κάποιος δεν τηρεί τα υπεσχημένα. Για να μην ξαναβρεθούμε σε μια κατάσταση που να είναι οριακή. Για να καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό το κοινό σχέδιο θα απαιτήσει εργαλεία για να μπορέσει να, να προχωρήσει, αλλιώς θα παραμείνουμε σε λίγο καιρό και πάλι σε μια κατάσταση παραομοία με αυτή της Λισαβόνας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και ο Πρόεδρος. Ο Γιώ Λάινεν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο τίτλος της στρατηγικής της Λισαβόνας ήταν η ανταγωνιστικότητα και ήταν μια μονομερής οικονομική στρατηγική η οποία εν μέρει απέτυχε. Είμαι ε, ε, πολύ ικανοποιημένος που ε, ο τίτλος της Στρατηγική Ευρώπη 2020 είναι η βιωσιμότητα. Αυτό είναι ο δρόμος που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Αποτελεί καλύτερη ισορροπία ανάμεσα ε, στην ε, οικονομική, κοινωνική και οικολογική ανάπτυξη και τις σχετικές ανάγκες. Η βιωσιμότητα έχει το μειονέκτημα ότι είναι μια ευρία έννοια, μπορεί να είναι και μια άδεια σακούλα. Θα πρέπει να την κάνουμε πιο συγκεκριμένη και το έγγραφο τη Κομισιόν είναι υπερβολικά ε, θολό για να μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Μια Ευρώπη με αποτελεσματικούς ε, πόρους, ε, αυτό είναι ε, πράγματι σωστό, διότι η ενέργεια και οι πρώτες ύλες μας δεν παρκούν. Ελπίζω μέχρι τον Ιούνιο να έχουμε πιο συγκεκριμένε προτάσεις ώστε να γνωρίζουμε τι θα πρέπει να κάνει ο καθένας, τι θα πρέπει να κάνει η Κομισιόν, τι θα πρέπει να κάνει το Κοινοβούλιο και τι θα πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη. Κάπως ξεχάστηκε ε, το θέμα του περιβάλλοντος ε, στην ε, Ευρώπη με αποτελεσματικούς πόρους, διότι έχει ξεχαστεί το θέμα. Θα ήθελα από την Επιτροπή Περιβάλλοντος περισσότερες οδηγίες σχετικά με το τι θέλουμε να κάνουμε. Η στρατηγική βιοπικιλότητα απέτυχε. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα μέχρι το 2020, θα πρέπει να συμπεριληφθεί και αυτό. Η προστασία του κλίματος ε, είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί πολύ. Πιστεύω ότι ε, θα πρέπει να στοχεύσουμε στο 30% και όχι στο 20% της μείωση ε, των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και ω προ την αποτελεσματικότητα τη ενέργεια είναι πολύ θολέ οι προτάσει, θα πρέπει να γίνουν δεσμευτικέ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Πιοτρόφσκι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η στρατηγική για το 2020 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι ιδεολογικής φύσεως. Η στόχη είναι αξιοπρεπής. Η αύξηση των το αριθμό των πτυχιούχων, ε, περισσότερα χρήματα για καινοτομία αλλά δεν προβλέπονται Ρώσεις για χώρες που δεν πετυχαίνουν τους στόχους. Θεωρεί κανείς ότι αυτοί που συνέταξαν τη στρατηγική δεν παρατήρησαν τη σοβαρή κρίση στην Ελλάδα και αύριο ενδεχομένω στην Ισπανία και την Πορτογαλία, κρίση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάρρευση της Ευρωζώνης και ενδεχομένω της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Μια τέτοια κρίσιμη στιγμή στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται λόγος για μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά 30%. Κάτι που θα πνίξει τις οικονομίες των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Πολωνίας συμπεριλαμβανομένης. Η πολιτική συνοχής επίσης κατευθύνεται προς προβλήματα. Η στρατηγική του 2020 είναι ουτοπικό σοσιαλιστικό πρόγραμμα. Ελπίζω να μην φέρει και άλλες ζημιές πριν καταλήξει εκεί που κατέληξε η στρατηγική της Λισαβόνας. Ευχαριστώ. Κυρία Χίμπνερ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για να είναι αποτελεσματική μια στρατηγική είναι απαραίτητο να δημιουργήσει δεσμούς μεταξύ στόχων και εργαλείων πολιτικής. Και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε ποιοι είναι οι μηχανισμοί που θα επιτύχουν τους στόχους της Ευρώπης 2020. Καταρχήν, ο κανονισμό τη εσωτερική αγορά που θα ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό και τον δυναμισμό τη ευρωπαϊκή αγορά και θα αναγνωρίσει τι κοινωνικέ υποχρεώσει που προκύπτουν από την οικονομική ολοκλήρωση. Θέλω να υποστηρίξω λοιπόν ιδιαίτερα αυτά που είπε ο Μάλκολμ Χάρμπορ. Δεύτερον, το θέμα τη επένδυση κεφαλαίου και η πρόοδο σε υποδομέ μεταφορών και τηλεπικοινωνών. Χρειαζόμαστε επενδύσει σε μια τεράστια πρωτοφανή κλίμακα. Τόσο οι δημόσιε όσο και οι ιδιωτικέ οι ε, επενδύσει θα πρέπει να κινητοποιηθούν και να υπάρξει συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Θα πρέπει τα ευρωπαϊκά πιστοτικά ιδρύματα να ενισχυθούν για να ξεπεράσουν τους ε, ε, φραγμούς που δημιούργησαν τα εθνικά έλλειμματα. Θα πρέπει επίσης μέσω από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό να υπάρξουν κοινέ δημόσιες δαπάνε, διότι μας ενδιαφέρουν κυριότερα τα θέματα τα οριζόντια και όχι ατομιακά. Γι' αυτό ο ευρωπαϊκός προπολογισμό θα πρέπει να βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη ε, προσέγγιση. Να ενισχύσουμε τα εργαλεία τα οποία θα οδηγήσουν στο άνοιγμα της οικονομίας μας στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Και εδώ απαιτείται και συνεργασία και συντονισμό σε επίπεδο εθνικών προϋπολογισμών μέσω της, εθνικής, της ε, λεγόμενης ενισχυμένης μεθόδου συνεργασίας. Όλα αυτά μπορούν να μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε στους στόχους του 2020, αλλά όχι μέχρι το στόχο. Είναι απλώς συνοδευτικά εργαλεία. Θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε περιοχές που μπορεί να προκύψει μια πραγματική ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία χωρίς να υποσκάψει τον ανταγωνισμό. Τα εργαλεία που έχουμε θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με ένα τέτοιο τρόπο ο οποίος δεν θα οδηγήσει σε μια ε, παρεμβατική κρατική λειτουργία η οποία θα υποσκάψει την ανταγωνιστικότητα σε διάφορους τομείς και αυτό θα μειώσει τη δυνατότητα ανάπτυξης της Ευρώπης και ο στόχος του 2020 πρέπει να είναι στόχος ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης δεν έχουμε καμία άλλη επιλογή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άρηφ για δύο λεφτά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση που διατρέχουμε είναι ανευπριγουμένου και πλήττει σκληρά την Ήπειρό μα και τον πληθυσμό τη, δημιουργεί τεράστιε δυσκολίε κοινωνικέ και ανθρώπινε και η Ελλάδα δυστυχώ είναι ένα παράδειγμα ομού και που βλέπουμε μπροστά μα. Η ανεργία συνεχώ αυξάνεται. Ήδη εκατομμύρια Ευρωπαίοι είναι χωρί απασχόληση και καθημερινά αυξάνεται ο αριθμό. Η απάντηση θα πρέπει να είναι πολιτική ισχυρή, γρήγορη, συντονισμένη, που θα λαμβάνει υπόψη τη σοβαρή περιβαλλοντική κρίση που ζούμε και που απαιτεί ένα νέο μοντέλο αναπτυξιακό. Αυτέ οι πολλαπλέ κρίσει δημιουργούν από την πλευρά των πολιτών μα μεγάλε προσδοκίε και ελπίδε στι οποίε η στρατηγική Ευρώπη του 2020 θα έπρεπε να απαντήσει. Αλλά είναι αυτών των προκλήσεων εξαιρετικού εύρου, η απάντηση δεν αντιστοιχεί και λυπούμε γι' αυτό. Οι προσανατολισμοί του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του περασμένου Μαρτίου δεν είναι στο ύψο των προκλήσεων, δεν υπάρχει φιλοδοξία, δεν υπάρχει βούληση, αλλά δυστυχώ αυτό δεν με εκπλήττει πλέον παντού εσείς οι ίδιοι μέλη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εσείς οι ίδιοι και η Επιτροπή σας ε, λέτε ότι έχει συνοχή πολιτικής. Έχω την εντύπωση, είναι πάρα ε, κάτι ένας, ε, που καλύπτει την έλλειψη δράσης. Ε, κοινωνική, οικονομική, εμπορική, πολιτική, βιομηχανική, γεωργική έρευνας δεν αναπτύσσονται για βιώσιμη ανάπτυξη και ισότιμη. Η εξωτερική δράση Ευρωπαϊκής Ενώσεω στην εμπορική πτυχή της είναι κάτι ανύπαρκτο. Ε, και νεοφιλελεύθερα δόγματα προς εκφράζονται. Θέλουμε το εμπόριο να είναι πραγματικά ένα εργαλείο για να δημιουργεί θέσει απασχόληση και ανάπτυξη, να καταπολεμά τη φτώχεια, να οδηγεί στην ανάπτυξη και δεν, να μην ακολουθείτε για τεχνικού λόγου, αλλά για λόγου πολιτικού και για διαφορετικού στόχου. Ε, θέλετε να μειώσετε το κόστο και και θέλετε συμφωνίε διμερεί. Ε, και όλα αυτά έχουν συνέπειε κοινωνικό ντάμπινγκ και φορολογικό ντάμπινγκ. Αυτέ οι πολιτικέ δημιούργησαν πάρα πολλού ε, που έχασαν τη δουλειά του, πολλέ μεταγκαταστάσει, πολλέ κοινωνικέ απώλειε. Λοιπόν, περιμένω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να ξαναδώσουν επνοή στο κοινωτικό πνεύμα, να αρνηθούν του εθνικού εγωισμού, ώστε η Ευρώπη να μην είναι μόνο μια, να έχει μια άβρα ευμαρία αλλά να δώσει και ελπίδα, να ανταποκριθεί στην εικόνα τη η Ευρώπη. Όχι μόνο εναντί των πολιτών τη, αλλά και του υπόλοιπου κόσμου. Αυτό είναι και το πνεύμα του ψηφίσματο ε, τη ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ. Ο κ. Ζέμπερ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ακούμε παρατηρήσεις των άκρων από δεξιά και από δεξιά δεν παίζουν ε, το ρόλο δυνάμεων που ενδιαφέρονται για την οικοδόμηση της Ευρώπης. Ε, ακούμε όμως ε, τη σύγκριση της Ευρώπης 2020 με πενταετές πρόβλημα του κομμουνισμού. Διαβάστε την ιστορία, θα καταλάβετε ποιες είναι οι διαφορές. Από την άλλη πλευρά Ε, και δεν εννοώ τις ε, φρόνιμες φωνές που, ε, που κάθονται εδώ ε, αμέσως στα αριστερά μας, αλλά όλοι ξέρουμε τι έχει προκύψει από την όλη κατάσταση. Πρέπει να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να επωφελούνται από την εκπαίδευση και τα άλλα αγαθά της κοινωνίας πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τους ε, υπάρχοντες πόρους. Το θέμα είναι ο προγραμματισμός. Οποιαδήποτε οικογένεια, οποιαδήποτε κοινότητα σκέφτεται τι μπορεί να κάνει με τους πόρους που έχει για να μπορέσει να προχωρήσει. Και νομίζω ότι είναι πολύ ε, σωστό να γίνεται κάτι τέτοιο. Μέχρι τώρα είχαμε μια ε, ε, ε, οικονομία αγοράς με ε, όρια. Δεν ήταν τελείως απελευθερωμένη. Θα ήταν φρόνιμο σε ευρωπαϊκό επίπεδο να σκεφτούμε την οικονομία αυτή της αγοράς, πώς μπορούμε να την οργανώσουμε στην Ευρώπη. Το να σκεφτόμαστε ε, ε, ε, εντό εθνικών ορίων δεν μπορεί να μας οδηγήσει στην επιτυχία πια. Πώς μπορεί η οικονομία αγοράς να εξυπηρετεί τους ανθρώπους. Το θέμα δεν είναι η ανταγωνιστικότητα αυτή καθεαυτή. Το θέμα είναι η Ευρώπη να είναι ανταγωνιστική ώστε να μπορούν να υποφεληθούν οι άνθρωποι. Ήδη πολλοί συνάδελφοι έχουν αναφερθεί στι λεπτομέρειε Εγώ θα ήθελα να περιοριστώ σε αυτή τη γενική παρατήρηση. Απλά θα ήθελα να πούμε στα κράτη-μέλη, σκεφτείτε τι θα κάνετε και πάνω απ' όλα διαβάστε την ιστορία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τικάο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως... Έχουμε φτάσει το 10% ανεργία στην Ευρώπη και 20% μεταξύ των ε, των ε, νέων ήταν πραγματικά θλιβερή η 1η Μαΐου γιατί η Ευρώπη έχει 23, 23 εκατομμύρια ανέργους. Για να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας θα πρέπει να δούμε σε ποιους τομείς θα πρέπει να επενδύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο με καλύτερη μόρφωση και κατάρτιση θα μπορέσουμε να δώσουμε στους νέους τις ε, απαραίτητες αξιότητες για να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους. Και οι επενδύσεις στη γεωργία θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια παραγωγή βασικών τροφιμικών προϊόντων και καυσίμων. Επίσης πρέπει να επενδύσουμε στις μεταφορές. Θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στα διευρωπαϊκά δίκτυα TEN-T. Χρειαζόμαστε τρένα υψηλής ταχύτητας που θα συνδέουν όλες τις ποτέβουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλες τις κύριες πόλεις, στις οποίες θα πρέπει να εξυγχρονιστεί η υποδομή του. Επίση, πρέπει να υπάρξουν επενδύσει στα λιμάνια, στι υποδομέ των μεταφορών, ιδίω στην Ευρωπαϊκή στην Ανατολική Ευρώπη και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ενιαία αγορά η οποία να είναι πραγματικά αποτελεσματική. Όλα αυτά απαιτούν δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία θα πρέπει να είναι η βάση που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και νέα έσοδα για τους ε, προϋπολογισμούς των κρατών μερών η ενεργειακή αποδοτικότητα και οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες ενέργειες θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, <clears throat> θα δημιουργήσουν 2,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας μέχρι το 2013. Όλα αυτά όμως χρειάζεται να γίνουν με επενδύσεις. Μα πάνω από 200 εκατομμύρια ε, χρημάτων τη στρατηγική ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν ακόμα επενδυθεί, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Θα ήθελα να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, ζητώντα από την Κομισιόν αλλά και από το Συμβούλιο να δημιουργήσουν ένα εργαλείο παρά, παρόμοιο με αυτό του Ταμείου Προσαρμογή στην, ε, στην παγκοσμιοποίηση για να αντιμετωπιστούν οι υπάλληλοι αυτοί που έχουν μείνει χωρί εργασία. Ευχαριστώ, κύριε Τζόρι. Ευχαριστώ Πρόεδρε olyan Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρετε ότι όλοι έχουμε ένα μεγάλο εγχείρημα ενώπιον μας. Χρειαζόμαστε μια πραγματική στρατηγική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι συνέπειε της κρίσης, αλλά επίση θα πρέπει να βρούμε και τον τρόπο να εξασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να ευδοκιμήσει και η οικονομία μας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε και τη δυνατότητα να δώσουμε στους πολίτες μας ένα υψηλότερο βιωτικό επίπεδο. Θέλω να πω δύο πράγματα. Γιατί η στρατηγική 2020 είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, ρεαλιστικοί και να θέσουμε εφικτούς στόχους, αλλά παρό... παράλληλα θα πρέπει να κατανοήσουμε και τις ιδιαιτερότητες των διαφορετικών κρατών μελών και τις διαφορές μεταξύ τους. Είναι κάτι διαφορετικό στο Ηνωμένο Βασίλειο η Ένδια από ό,τι στην Βουλγαρία. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτόμαστε αν θέλουμε να έχουμε 40% περισσότερους πτυχιούχους ή όχι στις χώρες μας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει μονάχα σε μεγαλύτερη ανεργία σε ορισμένε χώρες. Η δεύτερη παρατήρησή μου είναι η εξής. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να ενισχύσει την εσωτερική συνοχή και τη σύγκληση των οικονομιών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τους τομείς οι οποίοι είναι η λοκομοτίβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να μην ξεχάσουμε όμως ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές σε ό,τι αφορά το επίπεδο ανάπτυξης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να δώσουμε την πρέπουσα προσοχή σε αυτές τις διαφορές. Χωρίς εσωτερική συνοχή δεν μπορούμε να έχουμε ανταγωνιστικότητα προ τα έξω. Οι περιοχές οι οποίες έχουν υστέρηση ανάπτυξης θα πρέπει να τύχουν ειδικέ προστασίες, είναι οι μελλοντικέ αγορέ, είναι η μελλοντική ζήτηση για τα καινοτόμα προϊόντα και για αυτέ τι περιοχέ θα πρέπει να δημιουργηθούν τα κατάλληλα πλαίσια ώστε και αυτέ να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν την ενιαία αγορά, να γίνουν αυτόνομε και ανεξάρτητε και ανταγωνιστικέ και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια θέση αυτή τη νέα στρατηγική. Κυρία ή pirmininkė. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα μιλάμε για την διέρεση, για τις στόχους που θέτει σε 10 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα η ανεργία είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς αυτό μας κάνει να περιγράφουμε τη σημερινή νεολαία πολύ συχνά σαν τη χαμένη γενιά των σύγχρονων καιρών. Μιλάμε για την πρόθεση της πρωτοβουλίας για τους νέους, για την υποστήριξη των συστημάτων παιδείας και για άλλα σημαντικά στοιχεία. Όμως συνήθως μιλάμε για αυτά τα θέματα σαν μεμονωμένα και δεν βλέπουμε τη γενική εικόνα. Δυστυχώς όταν μιλάμε για τη στρατηγική για το 2020 μου δημιουργούνται ανησυχίες. Εγώ πιστεύω ότι θα παραμείνει ρητορικό σχήμα αν δεν ακούσουμε την άποψη των νέων. Ε, εκείνων που πρέπει να εφαρμόσει αυτή τη στρατηγική. Η στρατηγική το 2020 θα πρέπει να θεωρηθεί σαν συνεργασία μεταξύ οικολογία και οικονομία, ούτω ώστε οι νέοι να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τι γνώσει του και δεξιότητέ του για να δημιουργήσουν το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Εφόσον εκπροσωπώ εγώ την νεολαία, θα ήθελα να παρουσιάσω συγκεκριμένε προτάσει. Πρώτα απ' όλα, α υποστηρίξουμε τη δημιουργία των πράσινων θέσεων εργασία, όπω αποκαλούνται. Α ψάξουμε να βρούμε καλύτερου τρόπου για να υποστηρίξουμε τι επιχειρήσει που δημιουργούν πράσινη απασχόληση και απασχολούν νέου, είτε γεωργία, είτε στη βιομηχανία, είτε στι μεταφορέ, είτε στι υπηρεσίε. Δεύτερον, α δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στην προστασία του περιβάλλοντο και στην ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον. Αυτά τα δύο μέτρα από μόνα τους θα προσελκύσουν περισσότερους νέους στη δημιουργία ε, της πράσινης οικονομίας, της σύγχρονης οικονομίας. Εγώ θα ήθελα να ακούσω λιγότερους δισταγμούς και συγκρίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήθελα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, συγκέντρωση και αισιοδοξία. Ευχαριστώ. Και τώρα διαδικασία Catch the Eye. 19 συνάδελφοι έχω, έχουν ζητήσει το λόγο. Δεν μπορώ να βολέψω ούτε τους μισούς από εσά. Παρακαλώ να είστε υπομονετικοί. Ο κύριος Λούχαν έχει το λόγο. Για ένα λεπτό. Και ένα λεπτό, ε. Για να μιλήσουν και οι συνάδελφοί σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, αξιότιμοι συνάδελφοι, είμαι πεπισμένος ότι η Ευρώπη το 2020 θα είναι ισχυρότερη και πλέον καινοτόμα. Νομίζω ότι θα ξεπεράσουμε την κρίση διότι έχουμε τεράστιο δυναμικό όσον αφορά ε, την καινοτόμα εργατική δύναμη και τους πόρους και ε, εκτιμώ τις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά πρέπει να αναφέρω και την πολιτική συνοχής και θα ήθελα να εκφράσω την έλλειψη ικανοποίησή μου, διότι βλέπω ότι ο δρόμος προς τη Λισαβόνα φαίνεται να άλλαξε τελικά κατεύθυνση. Η κοινωνική και η τοπική συνοχή συνεπάγεται και άλλα πράγματα εκτός από ανάπτυξη ευφυή και ενταξιακή. Ε, οι πολίτες μας εξακολουθούν να λένε ότι χρειαζούνται υποδομές για τις υποδομές, για την πρόσβαση στις υπηρεσίες και την ανάπτυξη όλων των περιοχών ανεξάρτητα από το πόσο απομονωμένες είναι. Γι' αυτό το 2007 μέχρι το 2013 είδαμε ότι ετέθη, ε, υπογραμμίστηκε η σημασία των υποδομών και υποστήριξη της οικονομικής, του οικονομικού ανταγωνισμού για τη σύγκληση των περιοχών και η εξάρτηση μεταξύ πτυχών της οικονομίας καθιστά αυτό αναγκαίο. Η κυρία Ράπτη έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω συλληπιτήρια πρώτα από το βήμα αυτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στους τρεις συμπατριώτες μου που έπεσαν νεκροί σήμερα στα επεισόδια που είχαμε στην Αθήνα. Και λυπάμαι ειλικρινά που δεν άκουσα συλληπιτήρια εκ μέρους της κομισιόν από τον πρόεδρο μπαρόζο. ελπίζω ότι θα το κάνει στη δευτερολογία του ο κύριος Ρεν που τον εκπροσωπεί. το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να βιαστείτε στην επιτροπή. πρέπει να βιαστείτε γιατί όσο καθυστερείτε να δώσετε λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ευρώπη και άρα στο πρόβλημα της ελλάδας υπονομεύετε τους στόχους του. 2020. το 2020 βασίζεται στο 2010 ο στόχος να έχουμε λιγότερη φτώχεια βασίζεται στο σήμερα και με τα μέτρα που υποχρεούται να πάρει η ελλάδα δεν θα μπορέσει να συμβάλει σε αυτό το στόχο. υποχρεούστε να βοηθήσετε την ελλάδα γιατί διαφορετικά το 40% που πρέπει να είναι οι νέοι απόφοιτοι των πανεπιστημίων δεν θα έχουν δουλειά. σκεφτείτε το και βιαστείτε. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Μπαρόσο μίλησε για δράσεις τις οποίες θα πρέπει να αναλάβουμε στα πλαίσια της Ευρώπης 2020. Αλλά μετά εγκατέλειψε την αίθουσα και μία από τις ε, βασικές, βασικότερες δράσεις λείπει. Γι' αυτό ε, απευθύνομαι στην Ισπανική Προεδρία. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της ε, τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου που έχει παραμείνει εδώ πέρα και που ε, θα μπορέσει ε, να μας βοηθήσει. Ένα από τα βασικά ένας από τους βασικότερους στόχους είναι ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την βιώσιμη ανάπτυξη. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε το πράσινο δυναμικό και γι' αυτό χρειάζεται μια πρωτοβουλία για πράσινες θέσεις απασχόλησης. Και χρειάζεται μεταρρύθμιση. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα δικαιώματα των εργαζομένων ώστε να... και θα πρέπει να υπάρξει πρωτοβουλία για την ε, εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση. Ξέρω ότι η Ισπανική Προεδρία εργάζεται πάνω στο θέμα και ε, θα ήθελα να την υποστηρίξω. Ε, να του να το συνεχίσουν αυτό και να υποβάλουν πρόταση τη Προεδρία εντό του έτου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Thank um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συζητήσαμε για την Ευρώπη 2020, σε 10 χρόνια δηλαδή από σήμερα. Θα πρέπει όμως να σκεφτούμε τι έγινε τις τελευταίες 10 ώρες. Τρία άτομα σκοτώθηκαν, πέθαναν στην Ελλάδα. Θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες και τους οικείους τους, αλλά νομίζω ότι ξέραμε ότι θα υπήρχαν ταραχές, το είχα προειδοποίησει πριν από εβδομάδε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι καιρό στο Κοινοβούλιο μα, η Κομισιόν και το Συμβούλιο να ξυπνήσουν και να καταλάβουν ότι η Ευρωζώνη δεν λειτουργεί καλά. Είδαμε τα προβλήματα αυτά και τι τραχές στην Ελλάδα. Φοβάμαι ότι θα διαδοθούν προτού χαθούν και άλλε ζωέ, Ίσως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση των χωρών τη Ευρωζώνης και να, και να καταλάβουμε ότι υπήρξαν μεγάλα ασφάλματα στην κατασκευή του. Ο κ. έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθεί να είναι ισχυρότερη. Όμως, το Ελντοράντο μας αυτό δεν είναι αιώνιο. Οι κρίσεις, τα γεγονότα στην Ελλάδα δείχνουν τα κενά μας, τις ελλείψεις μας και θα πρέπει να μάθουμε το μάθημά μας. Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και αποφασιστικοί εφαρμόζοντας τη στρατηγική που ακολουθεί τη στρατηγική της Λισαβόνας. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι στο μέλλον ο κόσμος θα μπορεί να έχει το ίδιο επίπεδο διαβίωσης. Δεν είμαι σίγουρος όσον αφορά τους στόχους που έχουν τεθεί στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όταν 30% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν έχουν κανένα πτυχίο προσών. Θα πρέπει να είμαστε γρήγοροι και αποφασιστικοί. Όλοι οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι αποφασιστικοί στον φάτους στόχους της τη ε, παιδεία. Η κυρία Μπένοβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι κρίμα που δεν έμεινε ο πρόεδρος ε, της Κομισιόν. Ε, σίγουρα έχει σημαντικά πράγματα να κάνει, αλλά θα θεωρούσα ότι η ε, Ευρώπη 2020 είναι το πιο σημαντικό στρατηγικό υλικό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή επιτάπητος. Δεν μπορώ να φανταστώ τι πιο σημαντικό έχει να κάνει. Φοβάμαι ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 δεν έχει γίνει θετικά αποδεκτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κατάσταση στην Ευρώπη είναι δύσκολη και το έγγραφο έχει συνταχθεί με βάση μια από τις χειρότερες ε, οικονομικές κρίσεις ε, που έχει δει ποτέ η Ευρώπη. Η στρατηγική πρέπει να προστατεύσει τους πιο ευάλωτους ανθρώπους που ζούσαν ήδη υπό δύσκολες συνθήκες πριν την, κράση, πριν την κρίση, ε, που δεν φταίνε για την κρίση και που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Γι' αυτό θα έλεγα ότι Χρειάζεται η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός να συμπεριληφθούν στο διατακτικό του κειμένου. Δεν θα πρέπει απλά να αναφέρονται στο περιθώριο. Τέλος, η κυρία Μόρμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, το θέμα της, του μέλλοντος της Ευρώπης συνάπτεται με τη στρατηγική του 2020. Θα πρέπει να κατευθύνεται από δύο βασικές αξίες και οι οποίες συνδέονται ιδιαίτερα. Πρέπει να αγωνιστούμε για τις αξίες αυτές οι οποίες όμως δεν μπορούν να είναι παρούσες και ιδίως στην πραγματικότητα. Από τη μία μεριά έχουμε την παγκοσμιοποίηση και από την άλλη μεριά την βιωσιμότητα, την αηφορία. Δεν μπορούμε να ακολουθούμε και τις δύο. Ξέρουμε ότι η πορεία της παγκοσμιοποίησης είχε πολύ αρνητικά αποτελέσματα για το περιβάλλον και την αηφορία. και μπορούμε να μιλήσουμε και για την αηφορία στο κοινωνικό πλαίσιο, δηλαδή την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία είναι σημαντικά. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι τα θύματα του ανταγωνισμού, ανθρώπους οι οποίοι φτωχαίνουν όλο και περισσότερο και αυτό δεν μπορεί να ακολουθήσει την οδό της κοινωνικής αλληλεγγύης και αηφορίας. Πρέπει να μιζάρουμε στην αηφορία. Δίνω το λόγο στο Συμβούλιο στον κύριο Λόπες Γκαρίδο για να συνοψίσει την απάντηση του Συμβουλίου στα ερωτήματα που τέθηκαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριο Λόπες Γκαρίδο. Θα ξεκινήσω απαντώντας στο άμεσο ερώτημα το οποίο έθεσε ο κύριος Μπόκρος ο κ. Κομφεράτη αναφέρθηκε σε αυτό το ερώτημα που δεν είναι εδώ παρόν, όπω και η κυρία Δελκαστήγιο η οποία και αυτή δεν είναι παρούσα. Γιατί απέτυχε στατική τη Λισαβόνας είναι το ερώτημα. Αυτό είναι ένα σαφές ερώτημα το οποίο έθεσε άμεσα ο κύριος Μπόκρος. Λοιπόν, εδώ νομίζω ότι προφανώ είναι πολλοί οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την αποτυχία. Θα ήταν ίσω ε, φιλόδοξο μέχρι και αλαζονικό να θεωρήσω ότι του κατέχω όλου αυτού του λόγου. Αν έπρεπε όμως εγώ να επιλέξω κάποιο βασικό λόγο, κάποιο βασικό αίτιο, για μένα το πιο ουσιαστικό <clears throat> αίτιο που οδηγεί, οδήγησε στην αποτυχία της Αττικής Λισαβόνας είναι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ενέκρινε στο παρελθόν την ενιαία αγορά, ενέκρινε ένα ενιαίο νόμισμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έκανε το επόμενο βήμα που ήταν απαραίτητο για να επιτύχουμε την οικονομική ένωση. Δεν έγιναν τα απαραίτητα βήματα. Η συνθήκη του Μάστρι μιλούσε για οικονομική και νομισματική ένωση. Κάναμε την νομισματική ένωση, αλλά όχι την οικονομική. Δεν φτάσαμε ως εκεί. Γι' αυτό πιστεύω ότι μέσα στη στρατηγική 2020 θα πρέπει να εγγράψουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα νέο πλαίσιο που είναι η μετάβαση στην Οικονομική Ένωση η οποία σημαίνει πάνω απ' όλα μια κοινωνική και οικονομική διακυβέρνηση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα βασικό στοιχείο αυτής της οικονομικής ένωσης θα πρέπει να είναι μια στρατηγική ε, πλήρους απασχόλησης και δημιουργίας θέσεων εργασίας με ποιότητες. Αυτά είναι τα σημαντικότερα στοιχεία αυτής της ε, στρατηγικής για μένα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι παρεμβάσεις των βουλευτών, παρουσίασαν και νέα στοιχεία για την ε, στρατηγική αυτή. Το θέμα της τεχνολογίας, το θέμα της κοινωνικής στρατηγικής που ανέφερε ο κύριος Θέρκας και ο κύριος Κομφεράτη, ο κύριος Σαρίφ. Και επίσης η διάσταση του αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Και εγώ επανέρχομαι σε αυτά που είπε η κυρία Λάκα. Επομένως, δεν μπορούμε να επιτύχουμε χωρίς μια στρατηγική για θέσεις απασχόλησης ποιότητος και οικονομικής ανάπτυξης. Και αυτό το τόνισε και η κυρία Χάμς, η οποία δεν είναι παρούσα. Χρειάζεται κάτι το οποίο ανέφερε ο Επίτροπος Ολιρέν και το οποίο το επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή και θα το αναφέρει φαντάζομαι και στην επόμενη του ομιλία, την καλύτερη μορφή συντονισμού των κοινωνικών πολιτικών, πολιτικών απασχόληση και των οικονομικών πολιτικών στην Ευρώπη. Αυτό δεν έχει γίνει πραγματικότητα στην Ευρώπη και δεν το επέτυχε η στρατηγική τη Λισαβόνα. Η διαδικασία τη Λισαβόνα. Το άρθρο Πέντε τη συνθήκη της Λισαβόνας λέει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει, είναι υποχρεωμένα, πρέπει να συντονίζουν τις οικονομικές τους πολιτικές και τις πολιτικές τους απασχόλησης. Και εφόσον το επιθυμούν και πιστεύω πρέπει να το κάνουν, θα πρέπει να συντονίζουν και τις κοινωνικές τους πολιτικές. Πέραν της στρατηγικής αυτής απασχόλησης και πέραν του συντονισμού στον τομέα της απασχόλησης και της οικονομίας χρειάζεται μια ευρωπαϊκή εποπτεία των χρηματοοικονομικών αγορών. Αυτό είναι το πακέτο της εποπτείας, το οποίο γνωρίζετε και για το οποίο υπήρξε στο παρελθόν και η απάντηση του κ. Φερχόφστα, το οποίο στόνισε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό να εγκρίνει τη θέση του για το πακέτο χρηματοοικονομική εποπτεία. Επιπλέον, υπάρχει κάτι που ο πρόεδρο τη Κομισιόν, ο κ. Μπαρόσο, στην παρέμβασή του είχε υπογραμμίσει ιδιαίτερα. Θα πρέπει να υπάρχει και μια εξωτερική διάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να έχουμε μια ενιαία στάση εναντί του εξωκόσμου. Στους G20, παραδείγματος στις συνεδριάσεις αυτές. Και παραπέμπω σε αυτά που είπε ο πρόεδρος Μπαρός, που μπορώ να τις προσυπογράψω στο σύνολό τους. Χρειάζεται λοιπόν πέραν της Οικονομικής Ένωσης και τα απαραίτητα όργανα διακυβέρνησης. Ένα συμβούλιο το οποίο, ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο αναφέρει, το οποίο φασίζει βασικές πρωτοβουλίε Μια κομισιόν η οποία παρακολουθεί αυτή τη στρατηγική για το 2020 και δύο νομοθετικά όργανα, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και επίσης και κάποια εργαλεία για να δώσουμε θετικά κίνητρα προς την κατεύθυνση αυτής της στρατηγικής. Όπως είναι τα διαρθρωτικά ταμεία, τα οποία μπορούν να κατευθύνουν αυτή τη στρατηγική. Κάτι το οποίο δεν επέτυχε ιδιαίτερα για τα προηγούμενα χρόνια που ακολουθούσαμε τη στρατηγική της Λισαβόνης. Ε, εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά ήδη έχουν ξεκινήσει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρχίσει να κάνει το βήμα για την επόμενη φάση που απαιτεί η παγκοσμιοποίηση του 21ου αιώνα. Η Οικονομική Ένωση, όχι μόνο η εσωτερική αγορά, όχι μόνο η Νομισματική Ένωση, η Οικονομική Ένωση. Αυτή είναι η πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε με έναν τρόπο συνεκτικό, με διαθεσμικό διάλογο, όπως γίνεται σήμερα, και με τη μεγαλύτερη ταχύτητα αυτό μας ζητούν οι πολίτες της Ευρώπης σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Υπουργέ, τώρα ο Επίτροπος ο κύριος Ρέν θα πάρει το λόγο. Thank you, Madam President, Minister. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, κύριε Υπουργέ, ε, αξιότιμοι βουλευτές. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για ε, μια πολύ χρήσιμη συζήτηση απόψε. Επιτρέψτε μου να διορθώσω μια δήλωση σχετικά με τον πρόεδρο Μπαρόσο. Εξέφρασε την, τα συλληπιτήριά του στο όνομα της Επιτροπής. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου προς τις οικογένειες και ε, τους φίλους των θυμάτων της βίας ε, στην Αθήνα σήμερα. Η διαφωνία στην δημοκρατία είναι κάτι φυσιολογικό, αλλά το να προσφέρει κανείς τη βία δεν, είναι, δεν, μπορεί, να γίνει, δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε. Κυρίες και κύριοι, η βιώσιμη ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης βρίσκονται πράγματι στο, στην καρδιά της ε, Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Θα ήθελα να πω λίγα λόγια σχετικά με την χρηματοοικονομική σταθερότητα, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή στη βιώσιμη ανάπτυξη και στους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε Στατική Ευρώπη 2010, διότι πρέπει τώρα να ενεργήσουμε για να πετύχουμε ε, το 2020. Την προηγούμενη Κυριακή τα κράτη-μέλη αποφάσισαν ε, να κινητοποιήσουμε το ε, μέσο δημοσιονομικής στήριξης προς την Ελλάδα. Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη, ήταν όμως απαραίτητη. Ήταν μια υπεύθυνη απόφαση ήταν ε, αυτό που έπρεπε να γίνει. Έργο της Επιτροπής είναι τώρα να διασφαλίσει η ε, δημιουργική κινητοποίηση να ε, γίνει αποτελεσματικά και να εφαρμοστούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Η δημοσιονομική στήριξη προς την Ελλάδα της δίνει περιθώριο για να αποκαταστήσει την βιωσιμότητα των, ε, ε, δημοσίων, ε, των δημοσιονομικών αλλά και γενικά την ανταγωνιστικότητά της. Και είναι απαραίτητο αυτό όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά είναι απαραίτητο για να διασφαλίσει και την χρηματοοικονομική σταθερότητα στο σύνολο της Ευρώπης για να αποφύγουμε η πυρκαγιά στην Ελλάδα να εξαπλωθεί και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η οικονομική σταθερότητα είναι απαραίτητη για την ε, οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης, για την βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Κάποιοι από εσά αναφέρθηκαν ε, στη μεταδοτικότητα και τις ανησυχίες ε, για άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί ότι υπάρχουν εντάσεις στις χρηματαγορές τις τελευταίες μέρες και τις τελευταίες εβδομάδες αλλά πάντα στις ε, χρηματαγορές ε, βλέπουμε υπερβολικές αντιδράσεις. Τα κράτη-μέλη λαμβάνουν μέτρα για να σταθεροποιήσουν ε, τις οικονομίες τους, ιδιαίτερα η, Πολωνία, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Η Ελλάδα είναι ειδική περίπτωση στη ζώνη του ευρώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα η ζώνη του ευρώ, τα κράτη-μέλη μαζί με την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ε, έχουν αναλάβει την περίπτωση της Ελλάδας και ε, την υπόθεση της Ελλάδας ε, και είμαι πεπισμένος ότι θα πετύχουμε και θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις. Θα πρέπει να μάθουμε από την κρίση, αυτό είναι σημαντικό για την οικονομική διαχείριση της Ευρώπης ε, για το 2020. Οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρωπαϊκή οικονομία και ιδιαίτερα στην Ελλάδα και γύρω από αυτήν μας έχουν δείξει ότι υπάρχει επίγουσα ανάγκη να ενισχυθεί η δημοσιονομική διαχείριση στην Ευρώπη. Την επόμενη εβδομάδα η Κομισιόν θα υποβάλει συγκεκριμένε προτάσεις για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την, ε, το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ε, Οικονομική και Νομισματική Ένωση ε, το, ε, ε, ε, το νομισματικό ήταν πολύ πιο ισχυρό από το ευρωπαϊκό. θα πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν και την ευρωπαϊκή διάσταση. Αυτή άλλωστε ήταν και η ιδέα των ιδρυτών της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης. Η πρόληψη είναι πάντα πιο αποτελεσματική από τη θεραπεία και γι' αυτό θα πρέπει να βασίσουμε τις προτάσεις μας στην ενίσχυση της πρόληψης και ε, τον διορθωτικών μηχανισμών. Τα βασικά σημεία της πρότασής μας είναι τρία. Καταρχήν, θα πρέπει να ενισχύσουμε την σταθερότητα και το πακέτο ανάπτυξης ε, και όσον αφορά την πρόληψη και όσον αφορά τα διορθωτικά μέτρα. Χρειαζόμαστε πιο συστηματική ε, αλλά και έντονη εποπτεία των χρηματαγορών ώστε να αποφύγουμε στο μέλλον περιπτώσεις σαν αυτήν της Ελλάδας. Δεύτερον, θα πρέπει να ε, πάμε πέρα από την εποπτεία του υπολογισμού. θα πρέπει να ε, αντιμετωπίσουμε τις μακροοικονομικές ε, προκλήσεις και γι' αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε και την ανταγωνιστικότητα όσον αφορά τις εξαγωγές μας, κάτι το οποίο είναι επιγόντως απαραίτητο στα, σε πολλά κράτη-μέλη, αλλά και την εγχώρια ζήτηση θα πρέπει να την ενισχύσουμε όπου είναι απαραίτητο και όπου είναι δυνατόν. Το τρίτο στοιχείο είναι μηχανισμός επίλυσης της κρίσης. Ο οικονομικός μηχανισμός για την Ελλάδα ε, ε, ε, είναι απαραίτητο για την παρούσα φάση, αλλά είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε έναν μόνιμο μηχανισμό επίλυσης κρίσεων με ενσωματωμένες συγκεκριμένες προϋποθέσεις και αντικίνητρα για τη χρήση του. Ο πρόεδρος ε, Μπαρόσο είπε σήμερα ότι καλύτερα να ε, είναι κανείς προσεκτικός ε, παρά να μετανιώνει εκ των υστέρων. Θέλουμε να αποφύγουμε τα χειρότερα σενάρια στο μέλλον. Τέλος, κυρία Πρόεδρε, θα αξιότιμοι βουλευτές, στηρίζομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για, όσον αφορά την ενίσχυση της οικονομικής ε, διακυβέρνησης στην Ευρώπη. Καλό και τους αρχηγούς των κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξουν τις προτάσεις μας και να ενεργήσουν γρήγορα, χωρίς καθυστέρηση, στην υποβολή προτάσεων ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Γιατί, διότι δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου. Καλό όλους να λάβετε γρήγορα αποφάσεις ώστε η Ευρώπη 2020 να γίνει επιτυχία και να δημιουργήσουμε πραγματικές βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη. Αυτό περιμένουν από εμά οι πολίτες μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και για την αναφορά σας ε, στην κατάσταση στην Ελλάδα και τα αισθήματα που εκφράσατε αλληλεγγύης για τα θύματα σήμερα. Ε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στη διάρκεια της περίοδου συνόδου του Μαΐου 2 και τώρα θα ήθελα να σας ζητήσω να κάνουμε πέντε λεπτά διάλειμμα για τεχνικούς λόγους. Πέντε μόνο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ και θα συνεχίσουμε.